για να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 So, Αγαπητοί συνάδελφοι, θα συνεχίσουμε με τη συνεδρίαση της Επιτροπής μας. Φτάσαμε στο σημείο 20 της ημερήσιας διάταξης. Είναι το σημείο εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας για το Περιβάλλον. που αφορά τους νόμους και τα πρότυπα που ε, έχουμε συναποφασίσει εδώ. Μας ενδιαφέρει λοιπόν η εφαρμογή τους. Έχει έρθει η κυρία Πία Μπουτσέλα, που είναι διευθύντρια στη Γενική Διεύθυνση ΕΝΒΗ. Είναι υπεύθυνη για τις νομικές υποθέσεις και θα ήθελα να της δώσω το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Είμαι ευγνώμων και πολύ ευτυχής που βρίσκομαι εδώ, διότι για μία ακόμη φορά μας δίνεται την ευκαιρία να σας παρουσιάσουμε πώς εμείς προσπαθούμε να εφαρμόσουμε την κοινοτική νομοθεσία περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή. Είναι πολύ σημαντικό. Ίσως ο Επιτροπός μας ο κ. Γιάννα Ποτσόστιχ ε, κατά την ακρόασή του σα είπε ότι η εφαρμογή υπήρξε μία από τις σημαντικότερες προτεραιότητες του στη διάρκεια της θητείας του. Η Νέα Επιτροπή αναγνωρίζει τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε δημιουργώντας δύο υπηρεσίες και όχι πλέον μία. Αυτό λοιπόν είναι το πρώτο στοιχείο που θα ήθελα να υπογραμμίσω. Τώρα υπάρχουν δύο ξεχωριστές γενικές διευθύνσεις. Η Γενική Διεύθυνση του Περιβάλλοντος και η άλλη του Κλίματος. Και εμείς στη Γενική Διεύθυνση του Περιβάλλοντος θα δώσουμε ακόμη μεγαλύτερη σημασία από ότι ε, στο παρελθόν key sectors such as... σημαντικούς τομείς όπως η αντιμετώπιση των λιμάτων, ε, ε, των αποβλήτων και η αξιολόγηση εκτίμηση των επιπτώσεων. Αυτά, αυτοί είναι οι πυλώνες μας. Μία άλλη σημαντική εξέλιξη στη διάρκεια του περμένου χρόνου υπήρξε ε, ο διαχωρισμός των δύο νομικών υπηρεσιών μας και οι δύο ασχολούνται με τις παραβιάσεις η μία μονάδα έχει εξειδικευθεί όμως στο συντονισμό ε, της, των διαδικασιών αντιμετώπιση των παρελιάσεων και η άλλη μονάδα ε, έχει εξειδικευθεί ε, σε θέματα συμμόρφωσης ε, στη διακυβέρνηση. Αυτό υπήρξε δυνατό χάρη στην αύξηση του προσωπικού τα τελευταία χρόνια, κάτι που είχε ζητηθεί μεταξύ άλλων από σας και από ε, τους άλλους ευρωβουλευτές που συνεργάζονται μαζί σας. Αυτή τη στιγμή με υπερηφάνεια αναφέρω ότι καλύπτουμε σχεδόν όλες τις γλώσσες ε, των κρατών μελών. Θα ήθελα τώρα να σας μιλήσω για ζημένα θέματα, όπως ε, οι επιπτώσεις που έχει η συνθήκη της Λισαβόνας στο έργο που επιτελούμε και πώς θα προωθήσουμε την συμμόρφωση, πράγμα το οποίο ήδη κάνουμε, για συνεργαζόμενοι με ε, τους εθνικούς δικαστές σε θέματα περιβάλλοντος. Τώρα για τη συνθήκη της Λισαβόνας θα ήθελα να πω ότι η συνθήκη αυτή υπογραμμίζει δύο στοιχεία τα οποία είχαν περιληφθεί στην ανακοίνωσή μας του 2008 ότι δηλαδή οι παραβιάσεις θα πρέπει να αντιμετωπίζονται με ταχύτερο τρόπο. Η νέα συνθήκη επιτρέπει στην Επιτροπή σε περίπτωση όπου η μεταφορά στο εθνικό δίκαιο από τα κράτη-μέλη δεν γίνεται γρήγορα, ε, να ε, τους επιβάλλει πρόστιμα ήδη τη στιγμή που το δικαστήριο αποφαίνεται για πρώτη φορά. Αυτό είναι ένα σημαντικό νέο στοιχείο της συνθήκης. Επίσης, απαιτείται μόνο μία προειδοποιητική επιστολή σε περίπτωση κατά την οποία ένα κράτος μέλος δεν εφαρμόζει την δικαστική απόφαση. Συνεπώς, είναι ευκολότερο και πιο γρήγορο για την Επιτροπή να αποκτήσει, αν θέλετε, μια δεύτερη δικαστική απόφαση με επιβολή προστίμου, το οποίο όμως δεν σημαίνει ότι εμεί στην Επιτροπή ε, έχουμε ως αντικείμενο να επιβάλλουμε πρόστιμα στα κράτη-μέλη, ε, διότι ο χρόνος που απαιτείται για την αντιμετώπιση των παραβιάσεων δεν είναι τόσο μεγάλος όσο ο χρόνος και η ενέργεια που καταναλώνουμε όταν συνεργαζόμαστε με τα κράτη-μέλη για να επιτύχουμε τη συμμόρφωση για να επιτύχουμε μια σωστή εφαρμογή ε, της περιβαλλοντικής κοινωτικής νομοθεσίας εις όφελος ε, των πολιτών μας. Σχετικά με την πρόθεση της συμμόρφωσης στους κανόνες, καταρχήν αυτό που μας απασχολεί είναι η πρόληψη των παραβιάσεων. Ε, έχουμε πλατφόρμες συζητήσεων και ανταλλαγής απόψεων με τα κράτη-μέλη που αποτελούν ένα μόνιμο εργαλείο που μας επιτρέπει να εξετάζουμε μαζί τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν στην εφαρμογή της νομοθεσίας μας. Χρησιμοποιούμε scoreboards, πίνακες και πίνακες αποδόσεων. Αυτό είναι ένα στοιχείο που ήδη χρησιμοποιείται αρκετά χρόνια. Θα θυμάστε πόσο ισχυρό υπήρξε αυτό το εργαλείο των scoreboards όταν εισαγάγαμε το σύστημα ε, των γαλάζιων σημεών ε, για ε, τα ύδατα των λουωμένων στις θάλασσες. Επίσης οργανώσουμε διασκέψεις, εργαστήρια, σεμινάρια και επίσης ορισμένα έγγραφα καθοδήγησης που βοηθούν τα κράτη-μέλη να εφαρμόσουν καλύτερα την νομοθεσία μας. Επίσης, έχουμε σχέδια δράσης για την εφαρμογή των κανόνων, ώστε να βοηθήσουν τα κράτη-μέλη από την ημέρα όπου εσείς οι Ευρωβουλευτές ε, και το Συμβούλιο έχετε εγκρίνει μια νομοθεσία και να βοηθήσουμε τα κράτη-μέλη να εφαρμόσουν αυτή την νομοθεσία μέχρι την ημέρα όπου έχει πράγματι πραγματοποιηθεί, ε, εφαρμοστεί η νομοθεσία. Επίσης, πρόθεση των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο που βοηθάει τους πολίτες και τις μη να παίξουν σημαντικό ρόλο στην προστασία του περιβάλλοντος τους. Όπως γνωρίζετε, στον τομέα του περιβάλλοντος, η εργασία που επιτελείται από τους πολίτες, από τις ενώσεις πολιτών και από τις μη είναι κάτι το ιδιαίτερα σημαντικό για να υπάρξει γενική ευαισθητοποίηση των πολιτών στα θέματα του περιβάλλοντος και για να επιστήσουμε την προσοχή των κυβερνήσεών μας στην ανάγκη να βελτιώσουν την μεταφορά της κοινωνικής, την κοινωνικής νομοθεσίας του περιβάλλοντος. Πέρσι σε αυτό το τομέα εστιάσαμε στην μεταφορά των ε, δύο οδηγιών συμμετοχής ε, του κοινού. Οι πολίτες τώρα έχουν πρόσβαση ε, στους εθνικούς δικαστές και οι εθνικοί δικαστές πρέπει να είναι σε θέση να μπορούν να λειτουργούν πλήρως με βάση την κοινοτική περιβαλλοντική νομοθεσία. Έχουμε προς αυτή την κατεύθυνση ένα πρόγραμμα των ε, ε, ανταλλαγών βελτίστων πρακτικών ε, σε συζητήσεις με εθνικούς δικαστές ώστε να μπορούν να συζητούν μαζί μας και να ανταλλάσσουμε στοιχεία, πράγμα το οποίο μας βοηθάει στην εφαρμογή της κοινοτικής περιβαλλοντικής νομοθεσίας. Εδώ δεν πρέπει να λησμονούμε ότι οι εθνικοί δικαστές είναι κανονικοί κοινοτικοί δικαστές και συνεπώς ό,τι μπορούν να κάνουν οι εθνικοί δικαστές ε, δεν χρειάζεται να τεθεί υπόψη της Επιτροπής των Βρυξελών. Ήδη έχουμε ε, ε, δύο προγράμματα εκπαίδευσης των εθνικών δικαστών. Το ένα όσον αφορά την νομοθεσία σε θέματα της φύσης και την άλλη σε θέματα των αποβλήτων. Έχουμε μέχρι τώρα οργανώσει σεμινάρια στη Λιθουανία και στη Γαλλία και ε, θα λάβουν χώρα ε, την ερχόμενη εβδομάδα ακόμα τρία σεμινάρια στη Γερμανία, στη Σλοβενία και στο Ηνωμένο Βασίλειο και μετά το καλοκαίρι θα διοργανωθεί μια διάσκεψη στην Πορτογαλία όπου θα συμμετάσχουν οι Πορτογάλοι και οι Ισπανοί δικαστές. Αυτά τα ε, σεμινάρια κατέδειξαν ότι δεν υπάρχει μόνον ανάγκη αλλά και βούληση από πλευράς εθνικών δικαστών να συμμετάσχουν σε αυτές τις εμπειρίες. Αλλά βεβαίως δεν είναι πάντοτε δυνατόν να έχουμε ε, ένα καλό επίπεδο εφαρμογή ε, παροτρύνοντας μόνο τα κράτη-μέλη να κάνουν σωστά τη δουλειά τους. Συνεπώς, πρέπει να χρησιμοποιήσουμε όσο δυνατόν καλύτερα τον μηχανισμό εφαρμογής του νόμου που διαθέτουμε. Αυτή τη στιγμή εστιάζουμε σε τέσσερις τομείς προτεραιότητας όσον αφορά την εφαρμογή τη νομοθεσία, εκ των οποίων οι δύο υπογραμμίζονται, περιέχονται στις συνθήκες Λισαβόνα. Ο πρώτος τομέας είναι εκείνο που αφορά ε, την απουσία καθορισμού και εφαρμογή νομοθεσία επειδή δεν έχει γίνει η μεταφορά στην εθνική νομοθεσία. Ο δεύτερος τομέας αφορά τη μη συμμόρφωση στις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, Δηλαδή, όταν η πρώτη απόφαση δεν έχει εφαρμοστεί από ένα κράτος μέλος, τότε φτάνουμε στο τρίτο στοιχείο, το οποίο είναι ιδιαίτερα σημαντικό για μας και αφορά ε, ε, τα σημαντικά θέματα όπως η δημιουργία του ιστότοπου Natura και κατόπιν συστηματικές παραβιάσεις όπως το να ε, υπάρχουν παράνομες χωματερές ή η αδυναμία δημιουργίας κατάλληλων συστημάτων για το βιολογικό καθαρισμό των αστικών λιμάτων και επίσης οι παραβιάσεις σε μεγάλα έργα υποδομής. Και κυρίως αναφέρουμε εδώ στην αδυναμία ε, εκπόνησης ε, μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων ή να ληφθούν υπόψη ε, οι μελέτες που υπάρχουν. Λοιπόν, δίνουμε προτεραιότητα σε αυτές τις περιπτώσεις, διότι πιστεύουμε ότι αυτό ωφελεί τα μέγιστα ε, τους, περισσότερους πολίτες. Επίσης, έχουμε αρκετές υποθέσεις που αφορούν την έλλειψη περιβαλλοντικής υποδομής, όπως χωματερές και μονάδες βιολογικού καθαρισμού των αστικών λιμάτων. Ε, ένα άλλο παράδειγμα ήταν ε, το πρόβλημα των, αποβλήτων στην, ε, των απορριμμάτων στην Νότια Ιταλία το 2007 και την κρίση που ξέσπασε και ξεκινήσαμε, ενεργοποιήσαμε μια διαδικασία παραβιάσεων και ένα χρόνο μετά από την ενεργοποίηση αυτής της διαδικασίας Κάναμε προσφυγή στο δικαστήριο και θα ήθελα να σας πληροφορήσω ότι η απόφαση του δικαστηρίου αναμένεται ε, στις 4 Μαρτίου, δηλαδή προσεχώς. Επίσης, ασχοληθήκαμε με πολλά θέματα παραβιάσεων όσον αφορά την, ε, τον βιολογικό καθαρισμό των αστικών λιμάτων, διότι η έλλειψη βιολογικού καθαρισμού αστικών λιμάτων είναι το βασικό στοιχείο που δεν επιτρέπει την βελτίωση της ποιότητας των υδάτων σε όλη την Ευρώπη. Εδώ είμαστε αρκετά ικανοποιημένοι επειδή έχουμε αποκρίσεις από, από πολλά κράτη-μέλη όπως Βέλγιο, Ιταλία, Γαλλία, Πορτογαλία, Ισπανία και Ηνωμένο Βασίλειο. Φυσικά, για να δημιουργηθούν κατάλληλες μονάδες βιολογικού καθαρισμού, απαιτούνται μεγάλες επενδύσεις και χρόνος και για αυτό το λόγο παροτρύνουμε τα κράτη-μέλη να χρησιμοποιήσουμε ε, τα, τη χρηματοδότηση κοινότητας και έχουμε δημιουργήσει ένα χρονοδιάγραμμα, έχουμε καταρτήσει σχέδια δράσης, ώστε τα κράτη-μέλη να μπορούν να μας αναφέρουν σχετικά με ε, το στάδιο στο οποίο βρίσκονται ως προς την εφαρμογή των προγραμμάτων. Σε ορισμένε περιπτώσεις όμως υπήρξαν υπερβολικές καθυστερήσεις στην προετοιμασία αυτών των σχεδίων και δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο να χρειαστούν επιπλέον προσφυγές στο δικαστήριο και αντίστοιχη επιβολή ε, κυρώσεων και προστήμων. Αυτές, ως επιτοπλίστων, είναι οι περιπτώσεις έλλειψης των περιβαλλοντικών μελετών. Προσπαθούμε όμως ε, με αποτελεσματικό τρόπο και έγκαιρα να αντιμετωπίσουμε ε, και τα προβλήματα του, των πολιτών της Ευρώπης. Και εδώ προσπαθούμε να επιδείξουμε πνεύμα καινοτομία και χρησιμοποιούμε σε μεγάλο βαθμό ε, τα λεγόμενα πιλωτικά συστήματα που είναι ένα σύστημα γρήγορης απόκρισης που έχει δημιουργήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να μπορέσουν οι κυβερνήσεις και οι πολίτες που θίγονται να βρουν μια γρήγορη λύση σε ένα πρόβλημα. Φυσικά, όταν δεν προκύψει λύση μέσα στις προθεσμίες που έχουν τεθεί, τότε εμείς θα αναλάβουμε απευθεία την υπόθεση και επίσης σε ορισμένες πρωτεύουσες υπάρχουν συνάδελφοι που μας βοηθούν ως σύνδεσμοι με τη διοίκηση σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο και με τη βοήθεια των ΜΚΟ και των, πιλετών, και των πολιτών, ε, δίνουμε γρηγορότερες λύσεις στα προβλήματα από ό,τι θα κάναμε μόνοι μας από τις Βρυξέλλες. Θα ήθελα να καταλήξω λέγοντας ότι ναι, πράγματι, η Επιτροπή κατόρθωσε επιτελέσει σημαντική πρόοδο. Αλλά το περιβάλλον στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να μας επιτρέψει να εφησυχάσουμε. Υπάρχουν πολλές προκλήσεις που αντιμετωπίζονται σε τομείς όπως η διαχείριση των υδάτων, των αποβλήτων, ποιότητα ε, της ατμόσφαιρης και προστασία της φύσης. Και λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία αυτών των προκλήσεων, Είμαι πεπισμένη ότι το δικό σας το έργο ως Ευρωβουλευτών που ασχολείστε και στο επίπεδο της λήψης αποφάσεων αλλά και στο να μας παροτρύνετε εμάς την Επιτροπή να κάνουμε περισσότερα και να κάνουμε καλύτερα τη δουλειά μας στον τομέα της εφαρμογής Συνεπώς, η δουλειά που κάνει η Επιτροπή Περιβάλλοντος είναι πολύτιμη, επειδή μας επιτρέπει να φροντίσουμε ώστε πάντοτε οι φιλοδοξίες μας να, είναι, να βρίσκονται πολύ ψηλά για να εξασφαλίσουμε το καλύτερο δυνατό περιβάλλον για την Ευρώπη. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πουτσέλα για την παρουσίαση σας αυτή που έχει να κάνει με την εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας για το περιβάλλον. Πολύ ευχαρίστω ε, θα ανταποκριθούμε στην ε, έκκλησή σας ε, να συνεχίσουμε να πιέζουμε την Κομισιόν για εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας. Να την καλούμε να είναι φιλόδοξη στον τομέα αυτό, διότι τελείως δεν έχει νόημα να συναποφασίζουμε τους νόμους εάν η εφαρμογή δεν είναι ενιαία. Αυτός άλλωστε είναι ο στόχος του Ευρωπαϊκού Νομικού Χώρου. Ακούσαμε τι κάνετε για να πετύχετε την εφαρμογή του δικαίου στα 27 κράτη-μέλη. Μας αρέσει που ακούμε ότι η συνθήκη της Λισαβόνας αποτελεί πρόοδο στον τομέα αυτόν, ότι έτσι η εφαρμογή του περιβαλλοντικού δικαίου ε, μπορεί να οργανωθεί ώστε να πραγματοποιείται πιο γρήγορα. Ε, είπατε ότι οι διαδικασίες έχουν γίνει πιο σύντομες, ε, μπορούν να επιβληθούν πρόστιμα, τα οποία συνήθως πονάνε. Ό,τι δεν καταφέρνει κανείς ε, με λόγια, τα καταφέρνει με χρήματα. Μάλλον δεν έχετε κάνει κάτι τέτοιο ακόμα, διότι η συνθήκη της Λισαβόνας τέθηκε σε ισχύ 1η Δεκεμβρίου, αλλά ίσως μπορείτε στο τέλος να μας πείτε κάτι σχετικό. Είναι φυσικά σωστό να γίνεται συνεργασία με τα κράτη-μέλη, με τους φορείς, ε, προτού να καταλήξει κανείς σε ε, υποχρεωτικά μέτρα. Βρίσκω πολύ σωστά τα μέτρα ε, εκπαίδευσης των δικαστών, αλλά και η δουλειά που κάνετε στην διοίκηση σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Εργάζεστε, συνεργάζεστε και με την Επιτροπή των Περιφερειών. Ε, οι οποίε είναι υπεύθυνε ε, σε μεγάλο βαθμό για την εφαρμογή του δικαίου αυτού στα κράτη-μέλη. Βλέπω και που υπάρχουν τα προβλήματα. Η διάθεση των ε, απορριμμάτων, η προστασία του περιβάλλοντος είναι τα σημαντικά παραδείγματα όπου υπάρχουν σοβαρές ελλείψεις διαβάζοντας την ε, τελευταία έκθεση, την 26η από το έτος 2008, βλέπω ότι τα νούμερα είναι τρομακτικά. Στη σελίδα 4 λέτε ότι 55% της ε, ε, εφαρμογής που έπρεπε να γίνει το 2008 έχει καθυστερήσει. Βέβαια δεν είναι αυτό η επιτυχία που θέλουμε, απομένουν πολλά να γίνουν ακόμα. Εμείς πάντως θέλαμε έκθεση, δεν ξέρω αν κάποιος συνάδελφος έχει ερωτήσεις ή συστάσεις. Η Λίντα Μακέβαν. Μια ερώτηση για την Κομισιόν. Ευχαριστώ για αυτή την ε, πληροφόρηση. Στη συνθήκη της Λισαφώνας απαιτείται τώρα από εμά. Νομίζω, πρόεδρε, θα ήταν καλό καμιά φορά να έχει κανείς και μικρόφωνα μπροστά. Ξέρω ότι είναι θέμα πρωτοκόλλου, αλλά θα ήταν καλό να έχουμε μικρόφωνα μπροστά, ώστε να σας βλέπω κάστε, γιατί δεν γνωρίζω που είσαστε. Εκεί είσαστε δίπλα, ωραία. Λοιπόν, χρήσιμες πληροφορίες μας δώσατε. Γενικά στοιχεία, όχι συγκεκριμένα. Πάντως θα πρέπει τα εθνικά κοινοβούλια να δουλέψουν και θα το συστήσουμε στη συνέχεια. Αναρωτιέμαι όμω τι κάνει η Κομισιόν με τα Εθνικά Κοινοβούλια σε σχέση με το θέμα τη μεταφορά. Υποβάλλεται τίποτα στα Εθνικά Κοινοβούλια. Τα ενημερώνετε. Μπορούμε να το κοιτάξουμε αυτό το θέμα μελλοντικά. Επειδή και τα μέλη των Εθνικών Κοινοβουλίων θα πρέπει να ξέρουν ακριβώς πού αποτυγχάνει η μεταφορά. Και αυτό το ποσοστό 55% αποτυχίες μεταφοράς, τι γίνεται. Το αναθεωρούμε πριν εφαρμοστεί στις διάφορες χώρες. Δηλαδή πριν εφαρμοστεί ξεκινάμε αναθεώρηση να μην έχει ο κόσμος αυτή την ε, εντύπωση. Γιατί είχαμε αντίστοιχε περιπτώσει που αφορούσαν το Ηνωμένο Βασίλειο. Αναρωτιέμαι λοιπόν τι γίνεται εδώ με τα εθνικά κοινοβούλια, η καθυστερημένη εφαρμογή. Τι σημαίνει, σημαίνει ότι όταν θα κάνω μια θεώρηση νομοθετικής πράξης βρίσκουμε στη συνέχεια ότι οι μισές χώρες το κάνανε και ούτως ή συνεχίζεται δηλαδή επειδή αυτό ακριβώς το λέει στην νομοθεσία ότι πρέπει να το κάνετε ή τέλος πάντων έχετε πρόθεση, έχετε σκοπό να είστε πιο ευέλικτοι. Ευχαριστώ η κυρία Ροτμπέρετ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Η συζήτηση αυτή ε, είναι πολύ περίεργη κατά τη γνώμη μου. Έχουμε μια διαδικασία νομοθετική η οποία συνήθως διαρκεί δύο χρόνια με δύο αναγνώσεις. Ε, δεν είναι κακό αυτό. Τα δύο αυτά χρόνια έχουμε παράλληλα τις ομάδες εργασίας, ε, εργασίας του Συμβουλίου. Αποφασίζεται Υιοθετείται η νομοθεσία αυτή από όλα τα θεσμικά όργανα και βλέπουμε ότι τα κράτη-μέλη δεν θέλουν να την εφαρμόσουμε. Να, να τα εφαρμόσουν. Η κυρία Μπουτσέλα ε, είναι ευγενικό άνθρωπο και ε, βλέπει και την πλευρά των κρατών μελών. Αλλά εγώ δεν έχω τόση κατανόηση. Τα κράτη-μέλη θέλουν να καθυστερήσουν ε, την εφαρμογή με κάθε τίμημα. Ή λένε ότι είναι δύσκολο. Να, η Γερμανία έχει πολλά κρατήδια που δυσκολεύουν την κατάσταση. Άλλα κράτη-μέλη λένε ότι δεν ξέρουν λόγω της επιτροπολογίας δεν ξέρουν πώς πρέπει να γίνει. Ο απλός λόγος που μπορούμε να διαπιστώσουμε με νυφαλιότητα είναι ότι τα κράτη-μέλη δεν θέλουν να εφαρμόσουν την ευρωπαϊκή νομοθεσία και το βρίσκουν ενδιαφέρον. Την τελευταία εβδομάδα στο Στρασβούργο, όταν ε, επιβεβαιώσαμε την ε, νέα Κομισιόν, Υιοθετήσαμε ένα ψήφισμα το οποίο είχαμε διαπραγματευτεί με τον πρόεδρο της Επιτροπής Παρόσο, ε, που έχει να κάνει με μια νέα ε, διοργανική συμφωνία. Και μέρος της, του ψηφίσματος αυτού ήταν πιο γρήγορα να λαμβάνουμε πληροφορίες για τις διαδικασίες επί παραβάση, που αυτή τη στιγμή δεν λαμβάνουμε. Τις ε, λαμβάνουμε αργά, πολύ αργά, Αμέσως μετά, σε συνεδρίαση της Κορεπέρ, το Συμβούλιο τολμά να κάτσει να εξετάσει ε, εάν θα μας δώσει πληροφορίες σχετικά με το ποια κράτη-μέλη δεν εφαρμόζουν την νομοθεσία. Εγώ ανεπίσημα το έλαβα το έγγραφο αυτό, παράνομα, δεν, παρότι θα έπρεπε να λαμβάνουμε τέτοιες ε, πληροφορίες. τα κράτη-μέλη δεν θέλουν να δίνονται πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες επί Και είμαι πολύ αυστηρή στο θέμα αυτό. πολύ συχνά και το αναφέρατε κύριε Πρόεδρε, τόσο συχνά έχουμε προβλήματα με τα απορρίμματα, με την ποιότητα του νερού, με τη μόλυνση του αέρα. Τα κράτη-μέλη δεν εφαρμόζουν ή δεν ελέγχουν την εφαρμογή της νομοθεσίας. Η κυρία Μπουτσέλα είπε ότι θέλουμε να βοηθήσουμε τα κράτη-μέλη, να είμαστε παιδαγωγικοί. Ναι, αυτό το κάνουμε πριν ε, υιοθετήσουμε την νομοθεσία. Όταν την υιοθετήσουμε όμως ισχύει αυτή για 27 κράτη-μέλη με τον ίδιο τρόπο. Θα πρέπει λοιπόν να γίνει πιο γρήγορη η διαδικασία και κυρία Πουτσέλα θα ήθελα να μου πείτε το εξή. Ε, Πώ πιστεύετε ότι μπορεί να γίνει πιο γρήγορη η διαδικασία. Είναι πολύ απλά τα πράγματα. Η νομοθεσία θα πρέπει να εφαρμοστεί 1η Μαρτίου του 2010. Το πιο απλό πράγμα στον κόσμο είναι στις 15 ε, Μαρτίου του 2010 να λάβουμε από κάθε κράτος μέλος ε, μια επισκόπηση σχετικά με τον βαθμό στον οποίο έχει ε, εφαρμοστεί η νομοθεσία και αν όχι, γιατί όχι. Και εάν στις 15 Μαρτίου 2010 έχουμε την επισκόπηση αυτή, τότε θα πρέπει να στείλετε επιστολή σε κάθε κράτος μέλος που έχει καθυστερήσει. Παρακαλώ, στείλτε μας ε, μέχρι ε, την τάδε ημερομηνία τι έχετε εφαρμόσει. Ε, πινκ-πονγκ παίζουν εδώ πέρα, διότι λέμε, ωραία, έχετε δεν έχετε εφαρμόσει, τι δεν έχετε εφαρμόσει, γιατί δεν το έχετε εφαρμόσει. Και αυτό το πινκ-πονγκ συνεχίζεται επί 1,5 χρόνο. υπάρχουν ε, στην εποχή του email κάτι τέτοιο μπορεί να γίνει μέσα σε δύο εβδομάδες. Και έτσι, έξι μήνες μετά από την λήξη της προθεσμίας για εφαρμογή της ε, οδηγίας, ε, θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία αυτή. Ε, ναι, αυτό ήταν μια παρέμβαση όχι πολύ φιλική προς τα κράτη-μέλη, δίκαια θα μπορούσε να πει κανείς εφόσον υιοθετούμε ε, νομοθεσία την οποία δεν εφαρμόζουν και χάνουν χρόνο. Μέχρι να φτάσουμε στο, ε, στις διαδικασίες υπεραβάση συχνά περνάνε πολλά χρόνια και έχουμε συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης και εμένα θα με ενδιέφερε τη στιγμή που γνωρίζει κανείς μια ημερομηνία πώς μπορεί να εφαρμοστεί ένα τέτοιο σύστημα ε, έγκαιρης προειδοποίησης. Εάν έχουμε τώρα το 2010 και έχουμε μια προθεσμία μέχρι το 2011-2012, θα μπορούμε να ξέρουμε ποιος ε, τηρεί την προθεσμία και ποιο όχι. Συμφωνώ με, τον... με την Νομίζω ότι πολλές χώρες μέλη δεν θέλουν να τα εφαρμόσουν αυτά τα πράγματα και οι λόγοι συνήθως είναι θαυμάσιοι, αλλά δεν είναι συνήθως σωστοί. Εμεί δεν χρειάζεται λοιπόν να το αποδεχόμαστε αυτό θα πρέπει να επιταχυνθεί το, το χρονοδιάγραμμα. Ως βουλευτές βρισκόμαστε σε πίεση μεταξύ εθνικών κυβερνήσεων και των ψηφοφόρων μας που παραπονιούνται για αυτά τα πράγματα. Κάτι πρέπει να αλλάξει λοιπόν στην αρχή αυτού του θέματος πολύ και πολλές χώρες μέλη δηλαδή δεν θέλουν να τα εφαρμόσουν αυτά και κολυσιεργούν Πρέπει λοιπόν να έχουμε έναν τρόπο για να γνωρίζουμε ακριβώ ποιοι δεν κάνουν τα πράγματα που πρέπει να κάνουν επειδή θέλουν και ποιοι ενδεχομένω καθυστερούν επειδή αντιμετωπίζουν σοβαρού λόγου και δεν έχουν, έχουν δηλαδή σοβαρού λόγου να μην προσαρμοστούν σε ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Ευχαριστώ. Ο κύριο Τρομόπουλο. want to speak, you have to take the floor. Ε, ε, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, ήθελα να ε, ρωτήσω για ένα θέμα που αφορά την ε, Ελλάδα και την καταδίκη της ε, για, από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για την ύπαρξη χιλίων παράνομων χωματερών χώρων ανεξέλεκτης αναπόθεσης απορριμμάτων το 2005. Είναι ένα σοβαρό πρόβλημα και δεν έχει λυθεί. Ε, υπάρχει ε, κάποια άποψη ή προγραμματισμός για το πώς θα αντιμετωπιστεί το θέμα αυτό ε, και, εν πάση περιπτώσει, ποιες επιπτώσεις θα υπάρχουν λόγω αυτής της στάσης. Δεν έχει ζητήσει άλλο το λόγο η κυρία Πουτσέλα. Α, και η Άννα Ρόσπαχ ζήτησε το λόγο. Ναι, εντάξει, είναι αργά, αλλά δεν είναι υπερβολικά αργά για να ζήσετε το λόγο. Πολύ σύντομα θα ήθελα να ρωτήσω, μπορούμε να έχουμε κατάλογο των χωρών που δεν ελέγχουν ε, τα, τις παράνομες χωματερές τους. Ja, äh, vielleicht, wenn Sie da sagen, ob es so einen Anzeiger gibt. Äh, äh. Ναι, μήπως μπορείτε να μας πείτε ε, αν υπάρχει πίνακα σχετικά με την ε, τήρηση της νομοθεσίας ε, και της μη τήρησης της νομοθεσίας. Μπορείτε να μας πείτε ποιες χώρες είναι ιδιαίτερα αμελείς στο θέμα αυτό. Thank you. Ευχαριστώ για όλα τα σχόλια για όλα τα επικοδομητικά σχόλια. Θα ήθελα εγώ να προσπαθήσω να απαντήσω σε διαφορετικά σχόλια, δηλαδή για το ρόλο των Εθνικών Κοινοβουλίων και για το κατά πόσο η Κομισιόν βρίσκεται σε συζητήσεις με τα Εθνικά Κοινοβουλία. Πράγματι δεν είναι πολύ εύκολο για μας να έχουμε το χρόνο και την ευκαιρία να πάμε να μιλήσουμε σε κάθε Επιτροπή Περιβάλλοντος καθεσμιάς από τις 27 χώρες μέλη. Και μάλιστα η κοινοτική περιβαλλοντική νομοθεσία μεταφέρεται σε τοπικό περιφερειακό περιβάλλον. Οπότε θα έπρεπε να πάμε να μιλήσουμε σε ας πούμε 120 περιφερειακά κοινοβούλια. Ομολόγω ότι Εάν μας καλούσαν να μιλήσουμε σε κάποιο εθνικό κοινοβούλιο, ευχαρίστω θα το κάναμε. Όμως, σαν κανόνα δεν το κάνουμε αυτό. Παρ' όλα αυτά στο μέλλον, δεν αποκλείω τα ίδια τα εθνικά κοινοβούλια να δείξουν μεγαλύτερο ενδιαφέρον και λόγω της Λισαβόνας, εφαρμογής της συνθήκης Λισαβόνας, αλλά λόγω και του περισσότερο ευθύ ρόλου, άμεσου ρόλου που παίζουν τώρα τα Εθνικά Κοινοβούλια και στην εφαρμογή. Τώρα σχετικά με το κενό μεταξύ υιοθέτηση και εφαρμογής και για το τι κάνουμε. Εμείς στο παρελθόν παρατηρήσαμε ότι πολύ συχνά, εμείς ως Κομισιόν δηλαδή, θεωρήσαμε ότι όταν υιοθετείται μια νομοθεσία Πάει στις χώρες μέλη, επιστρέφει στις χώρες μέλη, όπου χρειάζεται αυτές να αναλάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για να εφαρμοστεί. Και επανερχόμαστε στην νομοθεσία αυτή όταν έχει εκπνεύσει η προθεσμία εφαρμογής. Βεβαίως αυτό να είναι και πολύ έτσι ενεργό ως δρόλος από την πλευρά της Κομισιόν και γι' αυτό ακριβώς τώρα έχουμε καθορίσει κάποια σχέδια μεταφοράς σε συνεργασία με τις χώρες μέλη όπου θα ελέγχουμε το μέχρι πού έχουν πάει οι χώρες στην εφαρμογή και για το κατά πόσο υπάρχουν κάποια κενά ή ελλείψεις που θα μπορούσαμε να αντιμετωπίσουμε. Και απατώντας την κυρία Ροτ να πω ότι πράγματι την ίδια μέρα όπου εκπνέει η ημερομηνία, η προθεσμία μεταφοράς και η γραμματεία της Κομισιόν δεν έχει λάβει τα μέτρα μεταφοράς από τις χώρες μέλη, τότε η νομική ε, δράση γίνεται αυτομάτως. Ξεκινά δηλαδή αμέσως, θα έλεγα, χωρίς καμιά καθυστέρηση και δεν χρειάζεται να γίνονται προεργασίες, ε, ερωταπαντήσεις, αλληλογραφία κτλ. Όχι. Η δράση αυτή ξεκινάει αμέσως και φτάνει μέχρι εκεί που χρειάζεται να φτάσει. Γιατί έχουμε διάφορες οριζόντιες διαδικασίες ε, παραβίασης και Πολύ συχνά οι χώρες μέλη αμέσως κάνουν τη μεταφορά λόγω αυτού του γεγονότος. Και βεβαίως ομολογώ έχουμε στη συνέχεια και το πρόβλημα του ελέγχου του κατά πόσο δηλαδή τα μέτρα για τη μεταφορά είναι σωστά. Αυτό είναι όμως ε, άλλο θέμα, τελείως διαφορετικό θέμα, γιατί πρέπει να δούμε και τη μεταφορά τι γίνεται σε περιφερειακό επίπεδο, κάτι το οποίο δηλαδή θα οδηγήσει σε πολλαπλασιασμό των μέτρων μεταφοράς και θα πρέπει και εκεί πάλι να ελέγξουμε κατά πόσο, και αυτό είναι και το χρέος μας, κατά πόσο τα μέτρα μεταφοράς είναι σύμφωνα με την κοινωτική νομοθεσία και εκεί έχετε δίκιο, χρειάζεται κάποιο χρονικό διάστημα, χρειάζεται κάποιος χρόνος. Η αλήθεια είναι ότι κάνουμε ό,τι μπορούμε, ό,τι είναι δυνατό, αλλά ίσως να μην κάνουμε το βέλτιστο, το καλύτερο και ευχαρίστως να παραδεχτώ ότι χρειάζεται χρόνος, όμως για την μη συμμόρφωση προχωράμε με τρόπο πολύ ευθύ και άμεσο. Δηλαδή ξεκινάμε αμέσως τη διαδικασία παραβίασης. Αυτό που ενδεχομένως ε, στέκει σε αυτό που λέτε είναι ότι αυτό το παιχνίδι τέλος πάντων υπάρχει το πινκ που αναφέρατε αλλά για τελείως διαφορετικό θέμα. Τώρα για την έλλειψη διαφάνειας σχετικά με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δηλαδή. Εμείς δεσμευόμαστε από τους τωρινούς κανόνες σχετικά με το τι μπορούμε να πούμε, τι μπορούμε να μεταβιβάσουμε, τι πρόσβαση στα έγγραφα μας δίδεται και προσπαθούμε λοιπόν να τηρήσουμε τους κανόνες όσο καλά γίνεται και τους τηρούμε, υπακούμε σε αυτούς τους κανόνες. Τώρα όμως είπαμε ότι όταν ξεκινάμε διαδικασία παραβίασης και όταν η παραβίαση είναι μια μεγάλη παραβίαση, τότε εμείς τίνουμε να εκδίδουμε ένα ανακοινωθέν τύπου για κάθε στάδιο της διαδικασίας παραβίασης. Γιατί συνοπτικά παρουσιάζει το ανακοινωθέν τύπου τα επιχειρήματα της Κομισιόν ενώπιον της κάθε χώρας μέλους και επιτρέπει και την κοινοποίηση, την δημοσιότητα αυτής της διαδικασίας δηλαδή παραβίασης. Θα έλεγα επίσης ότι εάν θέλετε να έχουμε ένα πίνακα βαθμολογίας. Οι πίνακες βαθμολογίας βρίσκονται καλύτερα στην ετήσια έκθεση, στις στατιστικές. Και η υπηρεσία περιβάλλοντος μας δημοσιεύει ετησίως στατιστικές σε σχέση με τις παραβιάσεις και αν κοιτάξει κανείς αυτές ακριβώς τις στατιστικές θα καταλάβει και θα δει πόσο γρήγορα ή αντιθέτως πόσο αργά προχωράμε στις υποθέσεις που αναλαμβάνουμε και πώς λειτουργεί το όλο σύστημα. Εγώ πάντως θα ήθελα να αναφέρω και πάλι αυτή την περίπτωση με τα απορρίμματα στην, νόμιο, νότια συγγνώμη, Ιταλία όπου πήγε στο δικαστήριο την Ιταλία η Κομισιόν σε λιγότερο από ένα χρόνο Παραπέμψαμε δηλαδή πολύ γρήγορα την Ιταλία στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για αυτή την υπόθεση και θα έχουμε την επόμενη εβδομάδα νομίζω και την τελική απόφαση του δικαστηρίου. Αυτό σε σχέση με τις δικές μας τις ε, πρακτικές ήταν πάρα πολύ ταχύ, ήταν πολύ γρήγορο σαν επίδεση. Τόσο γρήγορο λοιπόν, αυτό είναι το γρηγορότερο που μπορεί να τρέξει το σύστημα. Σε σχέση τώρα με τα τελικά ερωτήματα, με τελευταία ερώτηση για τα χαδά στην Ελλάδα, Νομίζω ότι είναι κλασική περίπτωση όπου η λύση προϋποθέτει μεγάλη χρηματοδότηση επειδή προϋποθέτει μεγάλη υποδομή, μεγάλες υποδομές. Και συγκεκριμένα σε αυτή την περίπτωση εμείς ενθαρρύναμε την Ελλάδα και η Ελλάδα το έπραξε να χρησιμοποιήσει τα ευρωπαϊκά περιφερειακά ταμεία ώστε να δημιουργήσει την υποδομή που χρειάζεται η Ελλάδα. Εμείς επιβλέπουμε την ε, πρόοδο όσον αφορά τη δημιουργία ενός νέου συστήματος διαχείρισης απορριμμάτων και το κλείσιμο των ε, χιτά στην Ελλάδα. Και αν δούμε ότι υπάρχει ανάγκη για άμεση δράση, αμέσως θα το κάνουμε. Προς το παρόν όμως, προς το παρόν όμως παρακολουθούμε στενά το χρονοδιάγραμμα το οποίο μας υπέβαλε η Ελλάδα ώστε να τηρείται αυτό. Αυτά, Πρόεδρε, προσπάσα να απαντήσω στις διάφορες ερωτήσεις. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Κυρία Πουτσέλα, θέλουμε να σας ενθαρρύνουμε να συνεχίσετε τη σημαντική αυτή εργασία, την εφαρμογή τον έλεγχο της εφαρμογής του περιβαλλοντικού δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σίγουρα θα επανέλθουμε στο θέμα αυτό και ελπίζουμε ότι θα έρθετε κι εσείς πάλι στην Επιτροπή μας ε, για να μας μιλήσετε για το επόμενο βήμα. Ευχαριστώ πολύ. Φτάνουμε στο θέμα 21 της ημερήσιας διάταξης. Αναδιατύπωση της οδηγίας ε, για τα απόβλητα ηλεκτρονικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Είναι πολύ ενδιαφέρον το θέμα αυτό. Ε. Το έχετε διαπιστώσει. Πολλοί επηρεάζονται από την νομοθεσία αυτή. Ε, η συγητής μας είναι ο Καρλ Χάινς Φλόρενς. Ε, έχουμε εδώ ένα πίνακα. Ήδη υπάρχει οδηγία από το 2003 τρεις χώρες έχουν μηδενική εφαρμογή μέχρι το τέλος του 2006, τρία χρόνια μετά δεν, έχουν κάνει τίποτα, δεν είχαν κάνει τίποτα μέχρι τότε. Υπάρχει λοιπόν ανάγκη ε, τη της οδηγίας αυτής. Ο Καρλ Χάινς Φλόρενς ε, έχει υποβάλει έκθεση και θα μας παρουσιάσει τώρα τις ιδέες ε, και τις σκέψεις του ε, σχετικά με το πώς μπορεί να βελτιωθεί η πρόταση της Κομισιόν. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Δεν συνεννοηθήκαμε με την Κομισιόν να συζητήσει σήμερα την εφαρμογή της ε, Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας για το περιβάλλον. Η οδηγία για τα απόλυτα ηλεκτρονικού και ηλεκτρικού εξοπλισμού είχε πολλά κενά. Το 2001-2002 διαμορφώθηκε η οδηγία αυτή ήταν ε, σαφές σε εμάς ότι δεν υπάρχει πουθενά στον κόσμο ε, ανάλογη ε, νομοθεσία και τα κράτη-μέλη ομόφωνα έλεγαν ότι δεν μπορούν, μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο, δεν θέλουμε να γίνει κάτι τέτοιο. Και έτσι είναι και σήμερα. Φαίνεται στην επισκόπηση ότι υπάρχουν χώρες, σημαντικές χώρες της Ένωσης, παλιές χώρες της Ένωσης, της Ένωσης των 15, έχουν μηδενική εφαρμογή ε, της οδηγίας αυτής. Είναι λοιπόν ε, καταστροφική εικόνα και κυρίως για το κοινοβούλιο μας, διότι τότε είχαμε καταβάλει σημαντικές προσπάθειες και τα κράτη-μέλη συμπεριλαμβανομένου του δικού μου κάναν ό,τι θέλουν. Θα πρέπει να σταματήσει αυτή. Αν υπάρχει λόγος ύπαρξης του κοινοβουλίου μας είναι να εφαρμόζονται αυτά που αποφασίζουμε μαζί με το Συμβούλιο. Αλλιώς ας πάμε σπίτι μας να κάνουμε κάτι άλλο. Γι' αυτό να πω σήμερα Α μην κάτσουμε να τσακωθούμε σήμερα αν θα μιλάμε για το 65% ή το 66%. Θα πρέπει να συνεργαστούν τα κράτη-μέλη. Κοιτάξτε, η Αυστρία. Η Αυστρία είναι πολύ ωραία χώρα. Σε γειτονική χώρα, εάν γίνεται ακριβώς το αντίθετο, τότε φανταστείτε ότι πολλά ε, πολλά ηλεκτρονικά απόβλητα θα μεταφέρονται στην ε, διπλανή χώρα. Ε, και αυτό είναι άδικο όχι μόνο για το περιβάλλον. αλλά και για την αίσθηση που έχουμε όλοι μας ότι δεν θέλουμε να εξάγουμε τα απόβλητά μας στις γειτονικές χώρες. Υπάρχει λοιπόν ένα σημαντικό θέμα εδώ πέρα και στην ε, οδηγία αυτή αλλά και στην οδηγία για την ε, διαχείριση των αποβλήτων. Υπάρχουν πολλά λάθη και θα πρέπει να κλείσουμε τα κενά ώστε να αξίζει ο κανονισμός ε, για την διαχείριση των αποβλήτων το όνομά του. Αυτό ήθελα να πω καταρχήν λοιπόν. από τα κράτη-μέλη θα ακούσετε ένα σωρό καλά επιχειρήματα. Για παράδειγμα ότι η καταχώρηση σε 27 κράτη-μέλη θα ότι η καταχώρηση θα πρέπει να γίνεται σε 27 κράτη-μέλη. Αλλά έχουμε μια ενιαία εσωτερική αγορά και προκαλεί έκπληξη ότι τα κράτη-μέλη μπορούν να πουλήσουν ηλεκτρονικό εξοπλισμό με 27 διαφορετικά ποσοστά ΦΠΑ. Αλλά όταν μιλάμε για την ε, συλλογή των αποβλήτων, ε, αυτό είναι πολύ δύσκολο και αυτό αντίκειται στις ε, βασικές αρχές της Ένωσής μας. Και η δική μου χώρα ασχολείται αυτή τη στιγμή με την διαχείριση των αποβλήτων ε, και θέλει να την, ε, να την κατευθύνει προς το εθνικό επίπεδο. Αυτό πονάει, αλλά... Προχωράμε προς την εξή ε, κατεύθυνση. Όταν κάποιος θέλει να δημιουργήσει ένα γλόμπο, θα πρέπει αυτός να μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε 27 κράτη-μέλη. Θα πρέπει λοιπόν να αλλάξουμε το σύστημα και ναι, δεν είναι απλό το σύστημα, αλλά δεν είναι όλα απαραίτητα αρμοδιότητα της ε, Κομισιόν. Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να εξετάσουν πώς μπορούν να καλύψουν το κόστος ενός ε, χρήσιμου και λογικού συστήματος ε, συλλογής ε, των αποβλήτων. Κυρίες και κύριοι, τα, τα ηλεκτρικά απόβλητα έχουν ραγδαία αύξηση έχουν αύξηση 150 τα 100 μέσα σε λίγα χρόνια ε, από ό,τι φαίνεται. Μέχρι το 2020 δηλαδή θα έχουμε τεράστια αύξηση. Ε, θα πρέπει να το φροντίσουμε αυτό. Το 2006 πουλήθηκαν ένα δισεκατομμύριο τηλέφωνα, το 2008 ήδη 1,8 δισεκατομμύρια κινητά. Σκεφτείτε ότι Σκεφτείτε ότι σε ένα εκατομμύριο κινητά υπάρχουν 250 κιλά άργυρος, 27 ε, χρυσό, 9 ε, κιλά παλάδιο. Ε, είναι πολύ χρήσιμα τα υλικά αυτά. Λοιπόν, θα πρέπει να... Ασχοληθούμε με την ανακύκλωση των τηλεφώνων αυτών. Θα πρέπει λοιπόν να σταματήσουμε και τις ε, παράνομες ε, μεταφορές των ε, αποβλήτων αυτών σε τρίτες χώρες. Διότι εκεί μπορούν να κάνουν πολύ μεγάλη ζημιά τα απόβλητα. Θα πρέπει λοιπόν τα κράτη-μέλη να αντιληφθούν τι ευθύνη έχουν. Μόνο αυτά μπορούν να διαπιστώσουν το ποσοστό που τελικά συλλέγεται. Κάποια κράτη-μέλη δεν θέλουν να ασχοληθούν ήδη με το θέμα, το αφήνουν αυτό στις επιχειρήσεις. Η Κομισιόν δεν μπορεί να απευθυνθεί στις μεγάλες επιχειρήσεις, Τα κράτη-μέλη πρέπει να ε, απευθυνθεί. Θα πρέπει όμως τα κράτη-μέλη να έχουν σαφείς κανόνες και στον κανονισμό για την ε, διάθεση των αποβλήτων ε, και στον, ε, και στον κανονισμό για τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Τα τελευταία δύο χρόνια έχει γίνει μελέτη, διαπιστώθηκε ότι από 400 κοντέινερ ε, που εξήχθηκαν και που ελέγχθηκαν, τα 380 ήταν παράνομα. 380 κοντέινερ από 400. Είχαν δηλωθεί τα κοντέινερ αυτά. Ε, ήταν ένα απλό κοντέινερ με απόβλητα. Ήταν κοντέινερ με απόβλητα αυτά, τα, ε, τα οποία απλά εξάγαμε εκτός Ευρώπης. Θα πρέπει λοιπόν όλοι να συμμετέχουν επί ίσης όρης στην ε, εφαρμογή ε, των κανόνων αυτών. Όλοι θα πρέπει να έχουμε... Όλοι ευθυνόμαστε για, για τον κακό έλεγχο των συνόρων και στην Σιγκαπούρη βρίσκουμε εκατοντάδες πλοία με ευρωπαϊκά απόβλητα που έχουν ε, εξαχθεί παράνομα. Αυτή λοιπόν η παράνομη εξαγωγή των αποβλήτων είναι σημαντικό πρόβλημα. Και με υψηλά ποσοστά, 25% προτείνει η Κομισιόν, θα πρέπει να ε, καταπολεμήσουμε το σύστημα. Πάντως, ε, σημαντικό είναι Υψηλέ υψηλές να οδηγήσουν σε έλεγχο από τα κράτη-μέλη. Φυσικά ελέγχουν τα κράτη-μέλη την κατάσταση, αλλά με πολλές ελλείψεις. Εδώ λοιπόν υπάρχει το σημαντικό πρόβλημα. Θα πρέπει να τονιστεί η ευθύνη των κρατών μελών στον τομέα του ελέγχου. Επίσης ε, σημαντικό είναι το υψηλό ποσοστό ε, συλλογής και θα πρέπει οι εξαγωγής να ε, να αποδεικνύουν ότι ο εξοπλισμός που εξάγουν λειτουργεί, διότι αν πρόκειται για απόβλητα, αν δεν λειτουργεί πια ο εξοπλισμός, τότε είναι παράνομη η εξαγωγή του. Τίθεται το θέμα των, κέντρων συγκέντρωσης, συλλογής ε, του υλικού αυτού. Υπάρχουν ε, διάφορες απόψεις για το θέμα αυτό. Στην ε, παλιά μας πρόταση προτείναμε οι Δήμοι να συλλέγουν τα υλικά αυτά και να πληρώνεται το σύστημα από τις επιχειρήσεις, διότι πιστεύω ότι καταναλωτής ενός ψυγείου ή ενός καταψύκτη έχει ευθύνη στον κόσμο τούτο. Ε, και ε, εάν, ε, εάν, εάν ο καταναλωτή απλά αρκεί να αφήσει το ψυγείο έξω από την πόρτα, τότε σε λίγο θα πρέπει να μπαίνουμε στο μπάνιο για να πάρουμε την παλιά του δοντόβουρτσα. Ε, αστεία το λέω, αλλά θα, έχει και ο καταναλωτή κάποια ευθύνη. Πιστεύω ότι θα πρέπει να υπάρχουν κέντρα συλλογή, δηλαδή στα οποία ο καταναλωτή να μεταφέρει ε, τον παλιό εξοπλισμό του. Εμένα στην πατρίδα μου όταν κανεί, κανείς δεν ήξερε τι είναι κέντρο συλλογής. Αν δεν το ξέρει κανείς αυτό δεν ξέρει πού να παραδώσει τον παλιό του εξοπλισμό. Θα πρέπει λοιπόν να εργαστούμε πάνω στο θέμα αυτό. Η Κομισιόν έχει ασχοληθεί με το θέμα του τι είναι το κέντρο συλλογή, ε, ποιο θα πρέπει να υποβάλει σχετικέ αναφορέ ε, και πώ μπορεί να γίνεται η διαπίστωση ότι έχει παραδοθεί ο εξοπλισμό στα ε, κέντρα συλλογή. Πάντω, διαπιστώνουμε ότι τα κράτη-μέλη δεν έχουν εφαρμόσει επαρκώ την νομοθεσία. Υπάρχουν πολλέ κατηγορίε και Ε, στην κοινωνία ακούει κανείς συχνά ότι έχουμε επιβάλει πολλή γραφειοκρατία. Ε, από 10 κατηγορίες εμείς ε, καταλήξαμε τελικά σε 5, διότι, διότι για κάθε κατηγορία θα πρέπει να υπάρχει σχετική γραφειοκρατική δομή. Έτσι λοιπόν, εγώ αντί για 10 κατηγορίες προτείνω 5 μικρές, ε, μικρό εξοπλισμό, μεγάλες, ε, μικρά, μικρές συσκευές, μεγάλες ε, συσκευές, γλόμπους κλπ. Υπήρχαν άλλοι που δεν θέλανε 10 κατηγορίες, θέλανε 15. Θα πρέπει να δούμε πώς θα προχωρήσουμε από εδώ. Είχαμε σημαντική συζήτηση σχετικά με τα τέλη. ο συνάδελφο Μπρέμ ήταν τότε, ήταν τότε ε, σκιώδης εισηγήτρια, το... έχει επανέλθει τώρα, ε, ε, εκείνη δεν ήθελε καθόλου να δεχτεί τα τέλη. Εάν δεν δεχτούν οι πολίτες να πληρώνουν τέτοια τέλη, τότε θα πρέπει να τα διαγράψουμε. Μπορεί κανείς να μιλάει για εθελοντικά τέλη. Όσον αφορά τα πρότυπα συλλογής και ανακύκλωσης, ε, Εδώ γράφω ότι η Κομισιόν θα πρέπει αλλού να θεσπίσει τους σχετικούς κανόνες, ε, όχι απαραίτητα σε τούτο το κανονισμό, αλλά αυτό κατά τη γνώμη μου δεν έχει γίνει ε, σε επαρκή βαθμό και κλείνω. Ε, θα ήθελα απλά να επαναλάβω ότι για μένα τουλάχιστον πρόκειται για αναδιατύπωση. Αυτό σημαίνει ότι επιτρέπεται να παρέμβουμε ως κοινοβούλιο μόνο στους τομείς όπου η Κομισιόν αποφασίζει ότι μπορούμε να παρέμβουμε. Εγώ έχω άλλη αίσθηση για τη δημοκρατία, αλλά εν πάση έτσι ρυθμίζεται το συγκεκριμένο θέμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οπότε φυσικά το δέχομαι. Ε, ό,τι είναι με γκρι στο κείμενο μπορούμε να το αλλάξουμε, τα υπόλοιπα δεν μπορούμε. Όσον αφορά το πεδίο εφαρμογή, αχ, μου, το ξέχασα αυτό. Δεν ξέρω. Γιατί Δεν, δεν ξέρω πώς έχει γίνει η ρύθμιση μέχρι τώρα ανάμεσα στο ΡΟΣ και το ΒΟΙ. είναι ο συγκεκριμένος ε, κανονισμός. Εν πάση πτώση, αυτά. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ, Καλ Χάινς Φλόρενς, για την ε, παρουσίαση του θέματος αυτού. Ανικανοποίητος ο Καλ Χάινς Φλόρενς με την εφαρμογή της οδηγίας. Οι σκιώδει εισηγητέ έχουν το λόγο. Κατλήν ehm, Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ επίση και τον εισηγητή. Ε, κύριε είμαι πάλι σιώδη εισηγητή, εισηγήτρια, δεν το είχα ζητήσει, αλλά μου το ζήτησαν. Και ίσω εν έχω γίνει πιο σοφή Ίσως εσείς το ζητήσατε, αλλά η έκθεσή σας πράγματι επιτελεί πρόοδο. Συμφωνώ ε, με το γεγονός ότι είναι τόσο φιλόδοξη αυτή η έκθεση, επειδή θέλετε να πείτε ότι η πρόταση δεν είναι αρκετά φιλόδοξη. Ε, και εγώ είμαι θυμωμένη από την περιορισμένη εφαρμογή της οδηγίας. Αλλά νομίζω ότι δεν, δεν, χρειάζεται να πω στην Επιτροπή ποιες είναι οι αξίες μας. Υπάρχουν πολλές προτάσεις που γίνονται από τον εισηγητή και δείχνουν την εκτίμηση της ομάδας μας. Ακόμα δεν έχουμε καταθέσει τροπολογίες, αλλά ευχαριστώ και τον συντονίστη. που έχει προβλέψει ότι ο φάκελος Austin Will θα αντιμετωπιστεί με την ίδια σοβαρότητα. Φυσικά όλα δεν θα είναι ίδια, αλλά τα δύο θέματα είναι αλληλένδετα. Συμφωνώ ότι πρέπει να έχουμε πάντοτε κατά νου τους μακρόπνους στόχους μας και προσωπικά αυτοί οι στόχοι αφορούν δύο τομείς. Δηλαδή, πώς μακροχρόνια μπορούμε να παροτρύνουμε τους παραγωγούς να ε, παράγουν προϊόντα ε, τα οποία θα σχεδιάζονται σωστά και με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και πώς να, θα φροντίσουμε να έχουμε όχι 60, 70, 80, 90% αυτών των προϊόντων. Αυτός πρέπει να είναι ο στόχος μας. Να συλλέγουμε αυτά τα προϊόντα όσο το δυνατόν περισσότερο. Τώρα, για το πεδίο εφαρμογής, Θέλετε να ανοίξετε αυτό το περιοριστικό κατάλογο της Επιτροπής όσον αφορά το παιδί εφαρμογή, συμφωνούμε, αλλά το ερώτημα είναι, χρειάζεται παρέκκληση για τις μεγάλες ε, σταθερές εγκαταστάσεις και τα ηλιακά πιάτα, διότι αυτό περιέχεται και στο φάκελο Ρώσο και αυτό γίνεται επειδή οι μεγάλες εγκαταστάσεις, οι σταθερές εγκαταστάσεις το απαιτούν, αλλά στην οδηγία για τα απόβλητα αναρωτιέμαι γιατί συμβαίνει. Επειδή μεγάλε σταθερέ εγκαταστάσει λόγω του μεγέθου του, λόγω του γεγονότο ότι είναι σταθερέ, δεν μετακινούνται και ακριβώ για αυτό το λόγο θα πρέπει ίσως να μας δώσουν κάποια εγγύηση οι κατασκευαστές. Αυτό είναι ερώτημα. Ως προς τον έλεγχο, νομίζω ότι πρέπει να μην έχουμε διαρροές, να αποφεύγουν διαρροές παντού, σε όλα τα σημεία. Επίσης, ο εισηγητής υπήρξε αρκετά απόλυτος, αλλά βεβαίως υπάρχει ευθύνη για τους παραγωγούς και θα πρέπει να προσδιορίσουμε αυτή την ευθύνη. Επειδή αυτοί οι οποίοι σχεδιάζουν τα προϊόντα, τα βγάζουν στην αγορά, θα πρέπει να φροντίσουν ώστε να επαναχρησιμοποιούνται αργότερα. Και αν δεν μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν, τουλάχιστον να γίνεται ανακύκλωση των προϊόντων αυτών 100%. Αυτή είναι ευθύνη των κατασκευαστών. Αν οι κατασκευαστές δεν μπορούν να καταστούν υπεύθυνοι για τη συλλογή, τότε ο καταναλωτής είναι εκείνος ο οποίος θα είναι υπεύθυνος. και τα κράτη-μέλη έχουν κάποιο ευθύνη, αλλά και οι καταναλωτέ. Αλλά δεν αρκεί να το λέμε. Πρέπει κάτι να κάνουμε. Σχετικά με την ευθύνη που έχει ο καταναλωτή. Ο εισηγητή κάνει μια πρόταση. Για να πλουστευθεί ο κατάλογος των κατηγοριών προϊόντων, ε, ναι, συμφωνώ να περιορίσουν σε πέντε αυτές οι κατηγορίες διότι έτσι η διαδικασία θα είναι πιο απλή, αλλά εδώ έρχομαι σε ένα πολύ σημαντικό σημείο, το οποίο θα συζητήσουμε ίσως διαμακρόν, ποιοι είναι οι στόχοι. Δηλαδή, τι θέλουμε να ανακτήσουν τα κράτη-μέλη σε αυτά τα απόβλητα των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών. Ποιο ποσοστό λοιπόν θα πρέπει να επαναχρησιμοποιηθεί, να ανακυκλωθεί. Αυτά είναι πολύ σημαντικά και πρέπει να γνωρίζουμε πολύ καλά τι είναι το ποσοστό που θέλουμε να ανακυκλωθεί. Ο Ευρωπαϊκό Οργανισμός Περιβάλλοντος, ε, οργανώσεις κατασκευαστών λένε ότι το 65% των προϊόντων που υπάρχουν στην αγορά θα πρέπει να ανακυκλώνεται. Νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει να βρούμε ε, κάποιον ορισμό και κάποιο στόχο. τα όσα έχουν, έχει κάνει και ο οργανισμός και οι κατασκευαστές είναι να βρεθεί ένα ποσοστό που ένα ποσοστό που θα είναι τα απόβλητα. Ώστε και πόσα μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν από αυτά τα προϊόντα. Αλλά αν δεν καθορίσετε στόχους ανά κατηγορία, Οπότε δεν ξέρουμε τι να κάνουμε. Δεν μιλάμε μόνο για υπολογιστές, για λάπτοπ κτλ. Αλλά και για τηλέφωνα, ακόμα και για ηλεκτρικές αποντόβουρτσες. Και θα πρέπει να βρεθεί ένα ποσοστό ε, των οικιακών συσκευών που θα πρέπει να επαναχρησιμοποιηθούν. Δεν πρέπει να τα πετάει κανείς στο δρόμο όλα αυτά τα μηχανήματα, τις συσκευές. Ε, υπάρχουν και τα κινητά τηλέφωνα, υπάρχουν μικροσυσκευές. Ακόμα, όπως είπα, και οι ηλεκτρικές οδοντόβουτσες που δεν τις ανακυκλώνει κανείς, τις πετάει στη σκουπίδια απλά και μόνο. Γι' αυτό, για να ανακτηθούν αυτά τα προϊόντα, πρέπει να προσδιοριστούν ποσοστά ανακύκλωση ανακατηγορία. το τέλος που θα καταβληθεί. Συμφωνώ με τα όσα είπε ο εισηγητής. Δηλαδή, θα πρέπει οπωσδήποτε να υπάρχει αυτό το τέλος και συμφωνώ ως προς την πρόταση που έκανε ο εισηγητής για τις εξαγωγές αντιστρέφει το βάρος απόδειξης και αυτό νομίζω ότι είναι σωστό. Πρέπει να ζητήσουμε να γίνονται περισσότεροι έλεγχοι. Σε μια βελγική εφημερίδα σήμερα αναφέρεται ότι αυτά τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά απόβλητα εξάγονται σε χώρες του τρίτου κόσμου από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από τι Ηνωμένε Πολιτείες αλλά και από χώρε όπω η Κίνα. Υπάρχει μια έκθεση του ΟΗΕ σχετικά. Λοιπόν, αυτές είναι βλαβερές για την υγεία και θα πρέπει να θέσουμε τέρμα. Ευχαριστώ, κύριε Στρομόπουλος. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Η αναθεώρηση της οδηγίας αυτής για τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού είναι μια σημαντική ευκαιρία για μια πιο αποτελεσματική τόνωση του οικολογικού σχεδιασμού των ε, σχετικών προϊόντων, για τη δημιουργία συνθήκων αντοχής στο χρόνο, ενάντια σε μια λογική που έχει κυριαρχήσει μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο για προσχεδιασμένη φθορά των προϊόντων, το οποίο είναι και ένα σημαντικό πρόβλημα. Δηλαδή είναι μια νέα μορφή εκμετάλλευσης όπου ενώ παλιότερα μια οικιακή συσκευή μπορούσε να κρατήσει μερικές δεκαετίες, να βγάλει τη ζωή ενός νοικοκυριού, έχουμε το φαινόμενο τα μεγάλα μυαλά στις διάφορες βιομηχανίες των ειδών που συζητάμε να σχεδιάζουν πόσο γρήγορα θα φθαρεί ούτως ώστε να αγοραστεί κάποιο καινούριο. Βεβαίως θα πρέπει να τονωθεί και η επαναχρησιμοποίηση και η ανακύκλωση και για να ενσωματωθεί το εξωτερικό κόστος στην τιμή των προϊόντων. Ζητήματα στα οποία είναι σαφές ότι η υφιστάμενη οδηγία δεν είναι ικανοποιητική. Μιλήσαμε για μια ευκαιρία. Για να μην περάσει αναξιοποίητη αυτή η ευκαιρία, η πρόταση της οδηγίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα πρέπει να βελτιωθεί ακόμη περισσότερο και να υπάρξει έμφαση στους παρακάτω τομείς. Την εξασφάλιση της εφαρμογής της αρχής της υπευθυνότητας των παραγωγών, ώστε αυτοί να καλύπτουν το πλήρες κόστος του κύκλου ζωής του εξοπλισμού. Ακόμη, την υιοθέτηση πιο συγκεκριμένων και φιλόδοξων στόχων συλλογής. Επίσης, την υιοθέτηση στόχου συγκεκριμένου για την επαναχρησιμοποίηση, καθώς επίσης και την αποφυγή διαρροών εξοπλισμού από την επίσημη και προβλεπόμενη αλυσίδα. Αν και η έκθεση Florence κάνει βήματα στην κατεύθυνση που περιγράφουμε, αρκετά ακόμη μένουν που πρέπει να συμπληρωθούν και να βελτιωθούν η έμφαση στην ευθύνη του καταναλωτή υποβαθμίζει τελικά το ρόλο των διανομέων και αγνοεί την ανάγκη για πόρους που έχει η αυτοδιοίκηση. Πιστεύουμε πως οι διανομείς θα πρέπει να εμπλακούν περισσότερο και πέρα από την πρακτική της ανταλλαγής της παλιάς με κάποια νέα συσκευή, για παράδειγμα μέσα από την απέτηση κάποιου ειδικού αποθηκευτικού χώρου ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού για διανομής ενός μεγέθους και άνω και την υποχρέωσή τους να λειτουργούν και ως σημείο συλλογής τουλάχιστον για τις μικρές συσκευές. Κάπου αυτό γίνεται. Ταυτόχρονα να απαιτηθεί από τα κράτη-μέλη να εξασφαλίσουν πόρους πάντα στη βάση της αρχής ο Ριπένον πληρώνει, να εξαφαλίσουν πόρους λοιπόν προς την αυτοδιοίκηση για εκστρατείες ευαισθητοποίησης της κοινή γνώμης και βελτιστοποίηση των ε, δημοτικών συστημάτων συλλογής. Θεωρούμε ακόμη σημαντικό να ενισχυθεί και να υποστηριχθεί η αποκομιδή εξοπλισμού από τα νοικοκυριά και όχι μόνο από τα σημεία συλλογής σχετικά με τους στόχους συλλογής. Η οδηγία θα ήταν πιο αποτελεσματική αν προέβλεπε συγκεκριμένους στόχους για επιμέρους κατηγορίες προϊόντων που είναι πιο πιθανό να οδηγηθούν σε ταφή όπως οι λαμπτήρες και οι μικρές συσκευές. Επίσης είναι σημαντικό να απαιτούνται πληροφορίες για τα παραγόμενα των μονάδων ανακύκλωσης και όχι μόνο για τις ποσότητες που στέλνονται για ανακύκλωση, τι γίνεται από εκεί και πέρα, προκειμένου να μετρούμε την πραγματική συνολική αποτελεσματικότητα του συστήματος. Σχετικά με την επαναχρησιμοποίηση, απουσιάζουν από την έκθεση αναφορές στην προτεραιότητα της επαναχρησιμοποίησης και της ανακύκλωσης σε σύγκριση με την καύση. Χρειαζόμαστε επομένω συγκεκριμένο και φιλόδοξο στόχο επαναχρησιμοποίησης, ενδεχομένως με δικαίωμα κατά προτεραιότητα πρόσβασης σε τέτοιους οργανισμούς. Σχετικά με την παρακολούθηση των ροών του εξοπλισμού και προκειμένου να παρακολουθείτε η αποτελεσματικότητα κάθε τμήματος της αλυσίδας, προτείνουμε τη συλλογή πληροφοριών εισόδου-εξόδου σε κάθε τέτοιο τμήμα. Επίσης, θα πρέπει να βελτιωθεί η παρακολούθηση των φορτίων του εξοπλισμού προς επιδιόρθωση και η παραγωγή αντίστοιχων αναφορών. Τέλος, το Ευρωκοινοβούλιο πιστεύουμε πως θα πρέπει να ζητά από όλα τα κράτη, όλα τα κράτη-μέλη υποχρεωτικά σχέδια βελτίωσης της διαχείρισης απορριμμάτων ηλεκτρονικού και ηλεκτρικού εξοπλισμού με αναφορά και αξιολόγησή τους προς την Επιτροπή. Ευχαριστώ. Äh. Ευχαριστώ πολύ. Κέρλινγκ. Ευχαριστώ. Να ευχαριστήσω για την έκθεση που παρακολούθησα με ενδιαφέρον. Υποστηρίζω τις αρχές της μεγιστοποίησης της συλλογή και ανάκτησης των πολύτιμων μετάλλων που χρησιμοποιούνται σε αυτά τα προϊόντα. Νομίζω όμως ότι ένα σωστό και κατάλληλο επίπεδο εφαρμογή οδηγία εδώ είναι απαραίτητο και αυτό που κοιτάμε εδώ είναι η αρχή τη ε, χρηστή νομοθεσία που είναι εύκολη να κατανοηθεί, ευκολονόητη, διαχείριστη και διευκολύνει και τη βιομηχανία. Σύμφωνα λοιπόν με αυτέ τι γραμμέ, νομίζω ο κύριο Φλόρεν και αυτή την αναζήτηση κάνει και αυτό ο ίδιο όπω λέγαμε προηγουμένω. Πάντως εμείς οι Ευρωπαίοι έχουμε κόλλημα με τα ηλεκτρονικά μας, συνεχίζουμε να τα αγοράζουμε, ακόμα τώρα και σε δύσκολους καιρούς συνεχίζουμε να κάνουμε αναβαθμίσεις και είμαστε προετοιμασμένοι να παρατήσουμε απόλυτα αποδεκτά προϊόντα προς χάρη της καινοτομία. Έχοντας λοιπόν υπόψη αυτή την στάση του καταναλωτή. Νομίζω ότι χρειάζεται να σκεφτούμε περισσότερο το πώ ο καταναλωτή θα συμπεριφερθεί και πώ θα μπορούσαμε να του δώσουμε κίνητρα και αυτό βεβαίω προποθέτει θα πρέπει να κατανοήσουμε περισσότερο νομίζω την αγορά στην οποία λειτουργούν. Γιατί στο τέλος θα μπορούσαμε να συζητήσουμε για τους παραγωγούς και την ευθύνη του Όμως, ε, στην ουσία ο καταναλωτή πληρώνει, είτε πληρώνει μέσω του κόστου του προϊόντος, είτε πληρώνει μέσω των φόρων, στι τοπικέ αρχέ, στι κυβερνήσει. με αυτού τους τρόπους δηλαδή. Εμείς πάντοτε πληρώνουμε. Πώς θα μπορούσε λοιπόν αυτό το κόστος ε, να μας βοηθήσει να ρυθμίσουμε αυτά τα θέματα. Εγώ δύσκολα βλέπω. Ίσως να υπάρχει κάποια φιλοδοξία εδώ. Αλλά δεν μας παρέχει τις απαραίτητες πρακτικές διαβεβαιώσεις για το πώς θα προχωρήσουμε. Πρέπει λοιπόν αυτό το συγκεκριμένο θέμα να το συζητήσουμε. Ε, όπως το θέμα και του πεδίου εφαρμογή. Το πεδίο εφαρμογή θα πρέπει να είναι ευθυγραμμισμένο με το πεδίο εφαρμογή των ρόλων μας που θέλουμε να έχουμε εδώ. Θα μπορούσαμε βεβαίως να το κάνουμε αυτό εν παραλίλω, αλλά νομίζω ότι θα είναι διοικητικά ανεξάρτητες αυτές οι προσπάθειες και ως ρόλους, αν δούμε το πεδίο, δεν έχουμε αποφασίσει ακόμα για το πεδίο εφαρμογή για το πώς θα είναι αυτό τελικά. Η άποψή μου είναι ότι δεν θα έπρεπε να είναι ανοιχτό, αλλά θα αλλάξει απλά και μόνο προς χάρη της αλλαγής. Εμείς πάντως θα πρέπει να αποφασίσουμε κατά πόσο να κάνουμε το ίδιο. Τώρα για τους στόχους, νομίζω ότι είναι σημαντική. Είναι σημαντικό να εξετάσουμε αυτά τα πρακτικά ζητήματα. Δεν προέχει μόνο η φιλοδοξία, αλλά και η πρακτικότητα. Το να μπορούμε να κάνουμε δηλαδή αυτό που θέλουμε να κάνουμε, γιατί είναι σαφές ότι δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Εντάξει, δεν φτάνει να είμαστε μόνο πιο φιλόδοξοι, αλλά πρέπει να είμαστε και πιο πρακτικοί. 65%, της, ε, ε, κανείς δεν νομίζω να διαφωνεί με αυτό το ποσοστό γιατί δίνουμε έμφαση στα βαριά προϊόντα και επιτρέπει στα μικρότερα προϊόντα τα οποία είναι πολύ πιο ανακτήσιμα από τους ε, καταναλωτές ή τέλος πάντων μάλλον είναι πιο εύκολα να αλλάχθουν από τους καταναλωτές οπότε δεν βλέπω λόγο να αλλάξει αυτό για τους ε, καταναλωτές, για τους μηνιαίους στόχους. Καταλαβαίνω τους στόχους αυτούς, αλλά νομίζω ότι θα έχει μεγάλο διοικητικό και γραφειοκρατικό φόρτο να γίνεται κάτι τέτοιο. Πολλές φορές μπορεί να αλλάξει ο καιρός ή δεν ξέρουμε πότε θα αλλάξει ο καιρός. Οπότε δεν ξέρουμε ακριβώς ας πούμε, πότε θα αγοράσει κανείς εξοπλισμό θέρμανσης ή κλιματισμού λοιπά, Οπότε είναι δύσκολο να ακολουθήσουμε αυτό το μηνιαίο στόχο. Μια αγορά για την οποία παραδέχεται ο κ. Λόιν στην ανάγκη συλλογής για ενέδος προϊόντων. Θα ήθελα εγώ εδώ να διευρύνουμε την κατηγορία αυτή, να είμαστε λεπτομερέστεροι και να δούμε το πώς ακριβώς αντιποκρίνονται μάλλον οι κατηγορίες σε σχέση με τους στόχους. Αν δεν το κάνουμε αυτό, δεν θα έχουμε τήρηση αυτών των στόχων μας εκ μέρους των καταναλωτών. Και τελικά νομίζω ότι αυτοί οι άνθρωποι, οι καταναλωτές δηλαδή, θα πρέπει να κάνουν αυτή τη δουλειά. Και θα πρέπει να τους οδηγήσουμε στο να κάνουν αυτή τη δουλειά. Τέλος δηλαδή, να πω και κάτι σε σχέση με το θέμα της, ε, της διαφανούς τιμολόγησης θα πρέπει να υπάρχει ένα έδος ορατής διαφανούς τιμολόγησης, όχι μόνο όσον αφορά την γέννηση του κάθε προϊόντος, αλλά θα πρέπει να υπάρχει και ένα έδος σημείωσης προς τον καταναλωτή ότι κοιτάξτε αυτό στοιχίζει κάποια χρήματα και ότι δεν το καταπίνει τελείω αυτό το κόστο στο κόστο του προϊόντο. Διαφορετικά θα αλλάξουν τη στάση του. Αν θέλουμε λοιπόν κάποιον πραγματικά να μπει στον κόπο, να ανακυκλώσει το κινητό του ή την ηλεκτρική βούρτσα, θα πρέπει να δώσουμε τα κατάλληλα κίνητρα να το κάνουμε αυτό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, η Σαμπίνε Βίλς. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να αφαιρθώ σε πέντε σημαντικά σημεία. Το ποσοστό συλλογής, ε, τα ποσοστά βάρους δηλαδή, ένα από τα σημαντικά σημεία του συναδέρφου Φλόρενς ε, είναι η η μέτρηση της ε, συλλογής ε, ε, κατά βάρος. Επίσης αναφέρεστε στην ανακύκλωση, αναφερθήκατε στις πρώτες ύλε που μπορούν να χαθούν και που θα πρέπει να αποφευχθεί, θα πρέπει να αποφευχθεί η απώλεια αυτή με την οδηγία αυτή. Η Οδηγεί αυτή θα χάσει την αποτελεσματικότητά της εάν έχει παραθυράκια. Πολύ συχνά οι μικρές συσκευές καταλήγουν στα κανονικά σκουπίδια. Εγώ πιστεύω ότι θα πρέπει να έχουμε αύξηση του ποσοστού συλλογής ε, και να γίνεται και χωρισμός σε κατηγορίες. Όσον αφορά την ε, καταχώρηση των κατασκευαστών ε, στα κράτη-μέλη, η διαλειτουργική, το διαλειτουργικό μητρό αποτελεί πρόβλημα καθότι οι επιχειρήσεις αυτές ε, δεν ε, ε, μπορούν να είναι υπόλογες στα άλλα κράτη-μέλη. Επίσης, δεν έχω καμία αντίρρηση σε ε, εθνική ενιαία καταχώρηση. Ιδιαίτερα οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις μπορούν να επωφεληθούν από αυτό. Τρίτον, όσον αφορά την ε, παρέκκληση για τα φωτοβολταϊκά, τα οποία περιέχουν κάδμιο. Αυτά δεν θα πρέπει να αποτελούν ε, παρέκκληση. Θα πρέπει ο στόχος ε, να είναι μετά από δύο χρόνια να αφαιρέσουμε από την παρέκκληση αυτή ε, οτιδήποτε περιέχει κάδμιο. Όσον αφορά την εξαγωγή παλιού εξοπλισμού, το καλό είναι ότι τώρα οι εξαγωγείς θα πρέπει να ε, αποδείξουν ότι ε, διατίθενται σωστά τα απορρίμματα αυτά, τα απόβλητα αυτά και είναι πολύ σημαντική αυτή η αντιστροφή του βάρους της απόδειξης. Ε, πρόβλημα παραμένει ωστόσο το ότι τα μεταχειρισμένα προϊόντα που εξάγονται αποδεικνύεται ότι λειτουργούν, εξάγονται λοιπόν, ε, χρησιμοποιούνται για κάνα δύο μήνες και μετά πάλι καταλήγουν στα ε, απορρίμματα. Όσον αφορά το πεδίο εφαρμογής, ε, συμφωνώ με την προσέγγιση του ανοιχτού πεδίου εφαρμογής να καλύπτονται δηλαδή όλες οι ηλεκτρικές συσκευές, ο δεσμευτικός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 Δεν ε, έχω φέρει μαζί μου έναν μακρύ τεχνικό κατάλογο, αλλά για μένα το σημαντικότερο είναι να ακολουθούμε τις βέλτιστες πρακτικές, διότι όπως το βλέπω εγώ το θέμα, το σημαντικό είναι ότι έχουμε 27 κράτη-μέλη με 27 διαφορετικές νομικές τάξεις. Από τους ανθρώπους που ασχολούνται με τις ηλεκτρικές συσκευές ακούω ότι Χαίρονται με την έκθεση του συναδέρφου Φλόρενς. Πιστεύω ότι θα ήταν καλή η ιδέα, αντί να έχουμε ένα σωρό τεχνικές λεπτομέρειες, να ρωτήσουμε τα κράτη-μέλη τι κάνετε τώρα. Δεν θέλω να τονίσω τη δική μου χώρα ως καλό παράδειγμα, αλλά είναι η χώρα που γνωρίζω καλύτερα και μπορώ να σας πω ότι στη χώρα μου έχουμε την εξής ρύθμιση. Έχουμε ε, κέντρα συλλογή στα οποία έρχεται ο ίδιος ο πολίτης ε, με τα μεγάλα του ε, απορρίμματα, τα οποία μπορεί να είναι οτιδήποτε, μπορεί να είναι πέτρες, και, να είναι μπάζα δηλαδή και να είναι, είναι μηχανές. Αυτό σημαίνει ότι ήδη ο πολίτης κάνει την, τον πρώτο διαχωρισμό των απορριμμάτων η προλαλή σας αναφέρθηκε ε, στα, ε, στον εξοπλισμό που ακόμα λειτουργεί. Μπορεί, ε, θα, μπορούσαν να υπάρχουν λοιπόν κέντρα όπου μπορεί να παραδώσει κανείς να μπορεί να πάει κανεί σε τον παλιό εξοπλισμό που λειτουργεί ακόμα σε κάποιο ειδικό κέντρο και κάποιο άλλο πολίτη να πάει να πάρει ένα μεταχειρισμένο, μια μεταχειρισμένη συσκευή που λειτουργεί ακόμα. Στη μικρή μου χώρα δεν γνωρίζω κανέναν που απλά να τα πετάει αυτά στα σκουπίδια του νοικοκυριού. Νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει να ακούσουμε ε, τι κάνουν οι διάφορες χώρες, να δούμε ποιες είναι οι βέλτιστες πρακτικές ε, και τι μπορούμε να κάνουμε για να καταφέρουμε ε, να κινητοποιήσουμε τον κάθε πολίτη στο θέμα αυτό. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ. Αυτή ήταν οι σκιώδεις εισηγητές. Ε, παρακαλώ τους επόμενους να μιλησουν δυο δύο-τρία λεπτά για να προλάβουμε. Ποιος θέλει το λόγο. Έχω πέντε που έχουν ζητήσει το λόγο. Ο κύριος Ρώση, η κυρία Κέρλινγκς. Εντάξει, να κλείσουμε το κατάλογο των ομιλητών. Η κυρία Μακίνας, παρακαλώ. Thank you, Chair. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, ευχαριστώ τον εισηγητή για την έκθεσή του. Νομίζω ότι καλή ιδέα είναι να δούμε τι λειτουργεί καλά σε ορισμένα κράτη-μέλη, ώστε να αντλήσουμε από την εμπειρία αυτών των κρατών. Το κράτο μέλο που γνωρίζω έχει δύο θέματα, τα οποία από ό,τι φαίνεται λειτουργούν. Πρώτα απ' όλα, ε, αυτό οι λιανοπολιτές τι πρέπει να πάρουν πίσω όσον αφορά με, ε, όταν... Ε, και αυτό λειτουργεί. Το δεύτερο, η δεύτερη ιδέα μάλλον που λειτουργεί, και ίσως δεν συμφωνήσουν προλαλήσαντες είναι αυτή, αυτό το τέλος, το ορατό τέλος όπως το λέμε. Νομίζω ότι αυτή η επιλογή ίσως καταστεί αναγκαία, διότι δείχνουν στους καταναλωτές ότι κάποια χρήματα πρέπει να πληρώσουν για να ανακυκλωθεί αυτή η συσκευή, ας πούμε, να την πάρουν πίσω. Και νομίζω ότι αυτό προβλέπεται εάν σε ένα κράτος μέλος ε, παρατηρήσουμε ότι αυτό έχει καλό αποτέλεσμα όσον αφορά τον όγκο των προϊόντων που ανακυκλώνονται. Η δυσκολία η δυσκολία εδώ είναι το εξή, ότι υπήρξαν πολλέ αντιδράσει. Τελικά όμω λειτουργήσε το σύστημα. διότι τότε είναι, είναι σαφέ ακριβώ ε, τι συμβαίνει. Αυτά τα δύο θέματα λειτουργήσαν σε εμά. Αλλά αν γίνουν αλλαγέ τώρα στο σύστημα το οποίο λειτουργεί, ε, θα υπάρξει κάποιο φόβο. Χρειάζεται αυτό το ορατό τέλο. Τώρα, για το πεδίο εφαρμογή, νομίζω ότι πρέπει να είναι ευρύτερο. Οι στόχοι είναι αναγκαίοι αλλά πρέπει να καθοριστούν καλύτερα λόγω των διαφορετικών μορφών συσκευών. Και επίσης ο διαχωρισμός σε πέντε κατηγορίες είναι μια καλή ιδέα. Αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε τελικά είναι να δούμε τι δούλεψε σωστά και ε, να τα εφαρμόσουμε. Αλλά όσο βλέπουμε πόσο περίπλοκο είναι το θέμα στην αγορά και ε, πόσε δυσκολίε υπάρχουν να προσπαθεί κανεί να νομοθετήσει ε, στα πλαίσια των διαφορετικών συστημάτων των κρατών μελών, Γι' αυτό νομίζω ότι αν υπάρχουν πολλέ λεπτομέρειε, το σύστημα θα είναι λιγότερο αποτελεσματικό. Επίση, οι τροπολογίε το δείχνουν. Πρέπει να αντλήσουμε στι ε, Καλέ εμπειρίε των κρατών μελών. Σε ορισμένε περιπτώσει, ε, ε, χώρε πραγματοποιούν το στόχο και το ξεπερνάνε. Νομίζω ότι αυτά τα καλά παραδείγματα πρέπει να τα ακολουθήσουμε για να αναμορφώσουμε την νομοθεσία μα και να πραγματοποιήσουμε του στόχου μα. Ευχαριστώ. Thank you very much, ε, Ευχαριστώ πολύ. Florence azt gondolom, Δεν ξέρω. Ε, πρέπει να πούμε ότι ο κ. Φλόρενς έκανε πολύ καλή δουλειά. Πάντοτε υπήρξε πολύ επιμελή στο καθήκον του. Θα ήθελα να υπογραμμίσω μια αντίφαση και έναν πιθανό κίνδυνο και θα ήθελα να κάνω ορισμένε προτάσεις για τροποποίηση. Πρώτα απ' όλα η αντίφαση. Η ανάλυση ότι θα πρέπει να έχουμε δηλαδή 65% συλλογή των ηλεκτρικών αποβλήτων. Με ε, τα 15 παλιότερα κράτη-μέλη θα το επιτύχουν το 2016. Και διαβάζουμε στο έγγραφο τα νέα κρατημέλη, τα 12 νέα κρατημέλη, το 2020 θα πρέπει να φτάσουν σε αυτό το στόχο. Εδώ υπάρχει μια αντίφαση. Παρά τα αυτά, παρόλα αυτά, παρά το γεγονός δηλαδή ότι ε, το έγγραφο για τους 12 αναφέρεται στο 2020. Το έγγραφο λέει ότι το 2016 οι παλιότερε χώρε έχουν επιτύχει το σκοπό του. Ε, Θα ήθελα τώρα να υπογραμμίσω ορισμένου κινδύνου. Ε, οι εμπειρογνώμονέ μου επέστησαν την προσοχή μου πάνω στου τυχόν κινδύνου. Μπορεί κάτι να αλλάξει με αυτό το έγγραφο. Παλιά μιλούσαμε για απομάκρυνση, τώρα μιλάμε για συλλογή. Η προηγούμενη λοιπόν έννοια εννοούσε ότι έπρεπε να απομακρύνουμε ε, αυτές τις συσκευέ με μηχανικό τρόπο. Ε, η νέα έννοια όμως προτιμάει τη χημική λύση. Αλλά εδώ υπάρχει ένα πρόβλημα όσον αφορά και την χρήση και την τεχνολογία. Ε, για παράδειγμα, στο παρελθόν μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε νοητικά καθυστερημένους για να κάνουν αυτή τη δουλειά. Αν όμως γίνει χημικά αυτή η δουλειά, αυτό σημαίνει ότι θα υπάρχουν λιγότερες πιθανότητες στα νοητικά καθυστερημένα άτομα να μπορούν να εργαστούν. Είναι ένα θέμα λοιπόν προστασίας του περιβάλλοντος, αλλά και θέμα απασχόλησης. Και είναι ένα θέμα κοινωνικής πολιτικής. Ε, αυτά είναι τα δύο σημεία από τα οποία θα ήθελα να ψήσω την προσοχή του κύριου Λόρενς. Ελπίζω ότι θα λυθούν ορισμένα αυτά τα προβλήματα. Ευχαριστώ. Θα πρέπει να ορίσουμε όμως ε, την συλλογή. Ο Βιτόριο Πρόντι έχει το λόγο. Ε, Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τον συνάδελφο Καλχάιντς για τη δουλειά του. Πρέπει όμως να ομολογήσω ότι αισθάνομαι κάπως άβολα μπροστά σε αυτή την ε, οδηγία, σε αυτή την πρόταση δηλαδή αναδιάμορφωσης και για το Ί και για το ΡΟΣ. Όπως ήδη είπαν κάποιοι συνάδελφοι, αυτές οι δύο οδηγίες θα πρέπει να συμπτυχθούν και θα πρέπει να αναδιοργανωθούν σύμφωνα με λειτουργικά κριτήρια θα έλεγα. Δηλαδή, εγώ βλέπω το Wii ως την οδηγία που θα πρέπει να στοχεύει στην ανάκτηση υλικών ή ολόκληρων τμήματων ή ανταλλακτικών αυτών των συσκευών που συσκευές σύμφωνα με τη φιλολογία είναι μακράς κατανάλωσης και ταχείας ανάκτησης. Εγώ λοιπόν εκλαμβάνω την ε, οδηγία WE ως αυτή που θα πρέπει να διασφαλίζει την ανάκτηση πολύτιμων φυσικών πόρων οι οποίες περιέχονται στις συσκευές χαλκός, ατσάλι, αλουμίνιο κλπ. Μετά τα σπάνια και πολύτιμα μέταλλα τα οποία βρίσκονται στα ηλεκτρονικά κυκλώματα και αυτά θα πρέπει να ανακτώνται. Εμείς λοιπόν θα πρέπει να σκεφτούμε την WE ως την οδηγία η οποία μας επιτρέπει να ανακτήσουμε οτιδήποτε μπορεί να ανακτηθεί και να αποφύγουμε ιδιαίτερα για τα σπάνια υλικά να αποφύγουμε λοιπόν μελλοντικές καταστάσεις ελήψεων γιατί αυτές ακριβώς οδηγούν σε συγκρούσεις. Επειδή λοιπόν αυτό συμβαίνει το ίδιο ισχύει και για τα υλικά το οποίο είναι το και τη ΔΡΟΣ. Γιατί αν ακριβώ είναι τμήματα ή ανταλλακτικά συσκευών, τότε θα πρέπει ή μηχανικού εξοπλισμού, τότε θα πρέπει να τα προσεγγίζουμε στο τελευταίο στάδιο ζωής της συσκευή. Ενδεχομένως λοιπόν θα μπορούσαμε να βρούμε έτσι μία διακλάδωση για τα πλαστικά παραδείγματι τα οποία χρησιμεύουν για πυροπροστασία θα μπορούσαμε να τα θέσουμε σε μια άλλη υποδηγία η οποία όμως θα πρέπει να πάει προς το reach το ταχύτερο δυνατό. Η διαφοροποίηση όμω σε αυτό ακριβώ το χρονικό σημείο θα πρέπει να γίνει. Και μάλιστα είναι αλήθεια ότι οι δύο οδηγίε, Ρίτ και Ρο, αναφέρονται στον ίδιο κατάλογο και στο ίδιο παράρτημα συσκευών. Οπότε εγώ δεν βλέπω νόημα να είναι χωριστές αυτές οι οδηγίες, οπότε σας ζητώ να το παναεξετάσετε και όπως έλεγα προηγουμένω με κριτήριο λειτουργικό, ώστε να αντιμετωπίζουμε από κοινού το τέλος ζωής της συσκευή, ώστε στη συνέχεια να διαφοροποιούμε ανάλογα με την ε, τοξικότητα και τις απαιτήσει που υπάρχουν εκεί. Θεωρώ λοιπόν ότι και για, τις, ε, και τα, για τα φωτοβολταϊκά είναι πολύ σημαντικό να γίνεται αυτή η διαφοροποίηση. Γιατί αυτή τη στιγμή ξεπουλιούνται τα φωτοβολταϊκά με γης 25 ετών και περιέχουν κάποια υλικά τα οποία είναι πάρα πολύ σημαντικά και τα οποία επιτρέπουν την, ανάκτηση. Κάδμιο επί και τελούριο. Το κάδμιο εντάξει είναι αρκετά μεγάλο σε ποσότητες, το τελούριο όμω. όχι. Οπότε αυτά θα πρέπει να μπορούμε να τα ανακτούμε ω υλικά. Να έχουμε λοιπόν υπόψη μας ότι το θέμα αυτό θα πρέπει να το μελετήσουμε σωστά και θα πρέπει να επικαλούμαστε το REACH επειδή εκεί ακριβώς θα πρέπει να ρυθμίζουμε τα θέματα της τοξικότητας. Όλα όμως τα υπόλοιπα θα πρέπει να αποβλέπουν κυρίως την ανάκτηση των υλικών. Αυτό ακριβώ θα πρέπει εμείς κατά νου και να θυμόμαστε ότι έχουμε να κάνουμε με καταστάσεις έλλειψης και τις οποίες θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε μελλοντικά. Το Wii λοιπόν θα πρέπει να αποτελεί μια ευκαιρία αντιμετώπισης αυτών των μελλοντικών καταστάσεων έλλειψης θα αντιμετωπίσουμε στο μέλλον. Ευχαριστώ. Ναι, είναι ενδιαφέρον το θέμα. Η συγχώνευση του ΡΟΣ και του Wii. Δεν θα πρέπει τουλάχιστον να υπάρχουν αντιφάσεις ανάμεσα στις δύο οδηγίες αυτές. Όσον αφορά τα φωτοβολταϊκά θα επανέλθουμε. Υπάρχουν ε, όμως ε, και άλλα προϊόντα τα οποία κρατάνε 20 χρόνια. Ωραίο το ότι τα φωτοβολταϊκά κρατάνε 20 χρόνια, αλλά υπάρχουν και άλλα τέτοια προϊόντα. Στην οδηγία ΡΟΣ θα πρέπει να δούμε λοιπόν σε τι βαθμό αυτό είναι προβληματικό. Θα πρέπει να γίνει σχετική συζήτηση. Ευχαριστώ πολύ. Ωραία Ρώση. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Να πω καταρχήν ότι συμφωνώ απόλυτα με αυτό που είπε ο συνάδελφο για την συγχώνευση οδηγιών Ράι που είπε ο κ. Πρόντι. Γιατί και εγώ θεωρώ ότι θα πρέπει να τα αντιμετωπίζουμε ως ενιαίο κείμενο ώστε να προλάβουμε μελλοντικέ καταστροφικέ καταστάσει. Τώρα, σχετικά με το κείμενο στο οποίο βρισκόμαστε τώρα, δηλαδή το ΡΑΕ, η αφιβολία που συνεχίζουμε να έχουμε και την οποία έχουμε αναφέρει είναι ότι το να φορτώσουμε όλε τι ευθύνε στι επιχειρήσει τη παραγωγή αυτό είναι λάθο γιατί σε πάρα πολλέ χώρε, όπω υπόθηκε σωστά και από τον εισηγητή, Υπάρχουν διάφορα κανάλια ανάκτησης των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών, τα οποία είναι ιδιωτικά και είναι από διάφορες μορφές. Δηλαδή το χαρίζουμε αν κάποιος έρθει να το παραλάβει κλπ. λοιπά. Υπάρχουν όμως κανάλια ανάκτησης ουσιώδη. Μετά τι γίνεται όμως με τις εταιρείες παραγωγούς που δεν έχουν την άδεια ανάκτηση. Ή θα πρέπει να κάνουμε νέους κανόνες συγκεκριμένου που υποχρεώνουν ένα κονσόρτσιουμ ανάκτηση. Δηλαδή όλους αυτούς οι οποίοι θα πρέπει να ασχοληθούμε αυτό το προϊόν ή αυτή τη συσκευή να κάνουν την ανάκτηση ή να δώσουμε δυνατότητα ανάκτησης σε, άλλες, σε άλλους φορείς. Κάτι το οποίο θα οδηγούσε σε φοβερές αυξήσεις του κόστους και βεβαίω αυτό στη τελική ανάλυση θα έχει επιπτώσει για τον καταναλωτή. Γιατί αν η επιχείρηση θα πρέπει να κυνηγάει τέλο πάντων τι διάφορε ροέ ε, για αυτή την ανάκτηση των συσκευών, αυτό έχει κόστο. Λογικό είναι λοιπόν η επιχείρηση να αυξήσει το κόστο αγορά για, τον, για τον καταναλωτή. Οπότε κάτι τέτοιο δεν γίνεται να το κάνουμε. Εξάλλου και το ποσοστό αυτό, 65% υποχρεωτικό ποσοστό ανάκτησης σε σχέση με το νεοπολιθέν προϊόν, αυτό είναι μια τρέλα. Γιατί αν παραδειγματικά μια χώρα ξεκινήσει ας πούμε μια εκστρατεία για τα παλιά αυτοκίνητα και δώσει τέλος πάντων κίνητρα για συγκεκριμένα είδη είτε αυτοκινήτων συσκευών γενικότερα δεν πειράζει, τότε σημαίνει ότι θα έχουμε μεγάλη αύξηση στις πωλήσει των συγκεκριμένων ειδών και αυτό θα είναι εις βάρος των υπολείπων συσκευών. Είναι δύσκολο λοιπόν να κάνουμε διαχείριση ποσοστιαία. Θα πρέπει να βρούμε μεθόδους πιο σωστές. Ευχαριστώ πολύ. Δεν νομίζω ότι ας πούμε για το eco-design. Οι συσκευές δεν νομίζω απαραίτητα να γίνονται ακριβότερες μελλοντικά. Ο επόμενος Το θέμα είναι σημαντικό και θα ήθελα να ξεκινήσω ευχαριστώντας τον συνάδελφο τον κύριο Φλόρενς για την πολύ καλή δουλειά που έχει κάνει σε, ένα, σε μια οδηγία που από τη φύση της είναι προβληματική. Ε, γιατί είναι προβληματική. Στην ουσία είναι προβληματική διότι ο καταναλωτής δεν έχει κίνητρο για να επιστρέψει πίσω την ηλεκτρονική συσκευή. Είναι υποχρεωμένοι η παραγωγή στην ουσία να κυνηγούν ε, όλο το σύστημα περιλαμβανομένων και των καταναλωτών. Οι παραγωγοί δικαίως παραπονιούνται ότι ένα μεγάλο κομμάτι του συστήματος λειτουργεί έξω από τις δικές τους δυνατότητες παρέμβασης και παρακολούθησης, περιλαμβανομένων και των παράνομων εξαγωγών, των πραγμάτων που πηγαίνουν από τους Δήμους οπουδήποτε αλλού κτλ. Και αυτό πρακτικά ε, σημαίνει ότι σε πάρα πολλές χώρες μέλη οι στόχοι αυτοί δεν επιτυχάνονται και αν θέλετε τη δική μου πρόβλεψη δεν πρόκειται και να επιτευχθούν. Όσο δεν αλλάζουμε την φιλοσοφία της οδηγίας γίνεται μια πρώτη προσπάθεια να αλλάξει φιλοσοφία και να μεταφερθεί ένα μεγάλο κομμάτι της ευθύνης στα κράτη-μέλη σε σχέση με τους παραγωγούς. Αυτό βεβαίως είναι μια ανακούφιση για τους παραγωγούς, αλλά δεν είμαι βέβαιος ότι είναι μια ανακούφιση για την ίδια την οδηγία. Δεν είμαι βέβαιος δηλαδή ότι τα κράτη-μέλη θα αποδειχθούν αποτελεσματικότερα από ότι η παραγωγή στην ε, προσπάθεια ε, αυτή. Ενδεχομένως θα πρέπει να αναζητήσουμε μία τρίτη λύση, μία ενδιάμεση λύση ή να σκεφτούμε περισσότερο δημιουργικά από ό,τι σκέφτηκε η Επιτροπή σε σχέση με τα κίνητρα που έχει ο καταναλωτής να επιστρέψει αυτές τις συσκευές, ιδίως σε σχέση με την σπάνη των αγαθών, όπως διατυπώθηκε από πολλούς συναδέλφους και βεβαίως έχουν δίκιο. Θα επανέλθω πάνω σε αυτό, απλώς να κάνω μία μικρή παρέμβαση για την υπόθεση των διανομέων. Οι διανομείς και ιδίω οι μεγάλοι διανομείς έχουν τις δυνατότητες να βοηθήσουν πολύ στην αύξηση του ποσοστού, διότι οι άνθρωποι όταν επισκέπτονται τους διανομής για να αγοράσουν μια καινούρια συσκευή, έχουν στο μυαλό τους την υπόθεση αγοράς και αν θέλετε και ε, από την προηγούμενη. Ενώ όταν βρίσκονται στο σπίτι τους αντιπέτωποι με, τον, ε, με την καθημερινότητά τους ή τον, το να κατεβάσουν τα σκουπίδια τους στο δρόμο, δεν έχουν την ίδια στάση, την ίδια αντίληψη. Οι μεγάλοι διανομής ιδίω από ένα μέγεθος και πέρα θα μπορούσαν να αναλάβουν μεγαλύτερο κομμάτι της ευθύνης για την συλλογή τουλάχιστον των μικρών ε, συσκευών και για τη διαμόρφωση μιας αντίστοιχης νοτροπίας του καταναλωτή. Αυτά ήθελα να πω και θα επανέλθω στο κομμάτι, στο θέμα κίνητρο στον καταναλωτή, γιατί ενδεχομένως να, υπάρχει και κάποιος, να υπάρχουν και άλλες ιδέες για να αυξήσουμε τα κίνητρα ε, επιστροφής αυτών των συσκευών. Ευχαριστώ. Ähm, να παρακαλέσω τον εκπρόσωπο της Κομισιόν να πάρει το λόγο πριν ο κύριος Φλόρινς κλείσει τη συζήτηση. Äh, äh, ναι, σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε που μας δίνετε το λόγο. Κύριε Σιγητά, κύριοι βουλευτές. First Το Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ Κοινοβούλιο λοιπόν και την Επιτροπή σας ιδιαίτερα για αυτή την ενδιαφέρουσα πρόταση και ευχαριστώ και τον εισηγητή βεβαίως για το σχέδιο στην γνωμοδότηση που συζητάμε σήμερα και το οποίο παρουσιάζει πάρα πολλά στοιχεία τα οποία συμπίπτουν με τη δική μας άποψη. Ξέρουμε ότι η οδηγία WE είναι σημαντική. Ένα από τα κρίσιμα ζητήματα μιας βιώσιμης παραγωγής και κατανάλωσης σημαίνει ότι ε, ανταποκρινόμαστε στους παραγωγού, στους καταναλωτές, τους αναφέραμε πολλές φορές απόψε και βεβαίως σημαίνει ότι εργαζόμαστε για μια κοινωνία ανακύκλωσης εδώ στην Ευρώπη και όχι μόνο. Και ιδιαίτερα αυτή η νομοθετική πράξη έτυχε παγκόσμια προσοχής και έχει χρησιμοποιηθεί και από άλλε χώρε ω καθοδήγηση για την πολιτική τους προσέγγιση σε αυτό το θέμα. Όλοι λοιπόν θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι το πρόβλημα WE, το οποίο ίσως αφορούσε την Ευρώπη, τη Βόρεια Αμερική και κάποιες άλλες χώρες υψηλού καταναλωτέ, είναι κάτι το οποίο αφορά όλο και περισσότερο τι αναπτυσσόμενε χώρε και τι αγορέ τους και τους καταναλωτές, καταναλωτές τους, οπότε αυτό θα πρέπει να μας οδηγεί ως παράδειγμα. Όπως ξέρετε, στόχος της οδηγίας είναι η επίτευξη του υψηλότερου δυνατού επίπεδου περιβαλλοντικής προστασίας. Και νομίζω ότι όλοι εδώ συμφωνούμε με την Κομισιόν ότι θα πρέπει να κοιτάξουμε τρία κυρία ζητήματα. Καταρχήν θα πρέπει να βελτιστοποιήσουμε την επεξεργασία του ΟΗ που έχει συλλεχθεί υπό την έννοια δηλαδή ότι θα πρέπει να υπάρχει η ελάχιστη δυνατή περιβαλλοντική επίπτωση και η μέγιστη δυνατή ανάκτηση. Δεύτερον, θα πρέπει να συλλέγουμε όσο we παράγουμε ώστε να ελέγχουμε και τον τελικό προορισμό του υλικού που συλλέγεται και αυτό φορά βεβαίω και τον γενικό προσανατολισμό της οδηγίας και τρίτον θα πρέπει να θέσουμε ένα παράδειγμα ιδιαίτερα σε εποχές όπως η δική μας να δώσουμε λοιπόν ένα παράδειγμα επίτευξης αυτού του υψηλού επίπεδου προστασία του περιβάλλοντο με όσο πιο αποτελεσματικό τρόπο γίνεται, χωρί βεβαίω να κάνουμε συμβιβασμού για την προστασία του περιβάλλοντο. Και η γνωμοδότηση του εισηγητή, κατά την άποψή μας, καθορίζει με τρόπο πολύ ξεκάθαρο αυτά τα τρία θέματα και από τα σχόλια που άκουσα σήμερα το απόγευμα όλοι νομίζω συμβαδίζουμε προς την κατεύθυνση αυτή. Επιτρέψτε μου μόνο για λίγα λεπτά να απαντήσω σε μεμονωμένα στοιχεία τα οποία αναφέρθηκα και ίσως να ήταν χρήσιμο να εξηγήσω το γιατί ε, πρότεινε αυτά που πρότεινε η Κομισιόν. Καταρχήν μεγάλο θέμα, το πρώτο μεγάλο θέμα σημαντικό, το πεδίο εφαρμογή. Βεβαίω λαμβάνουμε υπόψη μα την ευρύτερη υποστήριξη που τυχαίνει το ανοιχτό πεδίο εφαρμογή όχι μόνο εδώ στο σώμα αυτό, αλλά και σε άλλες χώρες μέλη. Θα ήθελα όμως για άλλη μια φορά να πω ότι θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί όχι με την υπερφιλοδοξία, αλλά με την βιασύνη ενδεχομένω εδώ. Γιατί κανένας από εμά δεν έχει μια σαφή εικόνα για το κόστος και το όφελος για το περιβάλλον που εμπλέκεται δηλαδή σε αυτή την κίνηση προς το ανοιχτό πεδίο εφαρμογής. Και αυτός μας, αυτό μας έκανε διστακτικούς και παραμένουμε διστακτικοί για να υποστηρίξουμε δηλαδή τη μετακίνηση προς ένα ανοιχτό πεδίο εφαρμογής χωρίς να έχουμε υπολογίσει σωστά το κόστος και το όφελος. Τώρα για το θέμα της ευθύνης, ποιος ήταν δηλαδή υπεύθυνο για την επίτευξη των φιλόδοξων στόχων συλλογής που έχουμε θέσει, η Κομισιόν στην πρότασή της, και αυτό το λέω επεξηγηματικά ε, για να σας βοηθήσει στη συζητήση σας, η Κομισιόν λοιπόν εδώ ακολούθησε την αρχή της ε, διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού στην λογική της επίπτωση δηλαδή. Εμείς εκτιμούμε, με άλλα λόγια, τα σχόλια τα οποία τονίζουν ότι η παραγωγή από μόνοι τους μπορεί να μην μπορούν να στηρίξουν την όλη προσπάθεια και θα πρέπει να χρειαστούν προσπάθειες και από άλλους φορείς και εμείς βεβαίως στην ίδια την πρόταση τονίσαμε αυτή την ανάγκη υποστήριξης εκ μέρους των ε, παραγωγών άρθρα 5 και 7 άρθρα 5 και 7 που παρουσιάζουν αυτό, αυτή ακριβώς την ανάγκη υποστήριξης εκ μέρους των χωρών μελών προς τους παραγωγούς αν αυτή τελικά η ευθύνη αποτελέσει τμήμα της ε, νομοθεσίας. Όταν μιλάμε στο ίδιο πλαίσιο για το να κάνουμε τους παραγωγούς υπεύθυνους για όλη την αλυσίδα συλλογής, δηλαδή από το σπίτι ξεκινώντας, η ιδέα πίσω από αυτή την πρόθεση, να σας εξηγήσω, είναι εξή ότι σήμερα η παραγωγή πληρώνει για οτιδήποτε συμβαίνει από τη στιγμή το φτάνει στο σημείο συλλογής. Και αυτό είναι δικό του κέρδος, δηλαδή τα απορρίμματα ανήκουν στους παραγωγούς και οτιδήποτε κέρδος προκύψει από, το, από τα απορρίμματα είναι δικό τους. Υπάρχει όμως και το θέμα της διαρροής εδώ, μεταξύ δηλαδή του, των οικειών και του ιδιωτικού σημείου συλλογής. Εκεί ακριβώς είδαμε δηλαδή ότι πολλά θέματα που αφορούν το γούι δεν λαμβάνονται υπόψη. Προσπαθήσαμε να καλύψουμε αυτό το κοινό, ανοίγοντας τη δυνατότητα και αφήνοντας δηλαδή τη δυνατότητα για τους παραγωγούς να καλύψουν σε αυτό το τμήμα της αλυσίδας από το σπίτι μέχρι το σημείο συλλογή, να λάβουν, μάλλον να καλύψουν το κομμάτι της οικονομικής ευθύνης από τη στιγμή βεβαίως που και τα υλικά που θα προκύψουν από την άκρη θα είναι δικά τους. Αναγνωρίζουμε βεβαίως ότι εδώ δεν γίνεται έχουμε μια νέα λύση μέσω της νομοθεσίας αυτής και όπως είδατε δεν προτείναμε ένα νομοθετικά δεσμευτικό κείμενο εδώ, απλά και μόνο μια σύσταση. Αλλά νομίζουμε ότι αξίζει τον κόπο να δούμε το πώς θα μπορούσαμε να αντιμετωπίσουμε αυτή την εφανή, τέλο πάντων διαρροή του WE. Το καταγραφή και αναφορά. Αυτά νομίζω ότι δεν θα θέλαμε να επιφέρει περιττό διοικητικό φόρτο στην οδηγία. Νομίζω ότι Αυτά που λέει ο εισηγητή ακολουθούν την ίδια κατεύθυνση με τις προθέσεις και τις ιδέες της Κομισιόν. Επί παραδείγματι το να αποφύγουμε το κόστος θέσπισης ενός ε, νομικού φορέα σε 27 χώρε, ή σε ξέρει πόσε πόσες άλλες χώρες ακόμα. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα σημαντικό βήμα αποφυγής περί του φόρτου το οποίο σημαίνει ότι η ίδια διοίκηση θα πρέπει να είναι υπεύθυνη και βεβαίω και χρησιμοποιεί και όλα τα μέσα όπω τα ηλεκτρονικά μέσα ε, για την διευθύνση αυτού του θέματο και αυτό είναι η ίδια ιδέα που έχουμε και εμεί. Τώρα το λογικό αντίτιμο το αναφέρατε πολλοί από εσά και το αναφέρατε ενδεχομένω και ω επίμαχο ζήτημα. Γιατί η Κομισιόν λοιπόν προτείνει να διατηρήσουμε αυτό το ορατό, το ξεκάθαρο ή ευκρινές τέλο πάντων τίμημα. Εμείς θέλουμε να πάμε από την κατανάλωση στην βιώσιμη κατανάλωση και θεωρώ ότι υπάρχει ευρεία συνένεση για το γεγονό ότι στόχος της βιώσιμης κατάστασης, κατανάλωση συγγνώμη, είναι η ενημέρωση των καταναλωτών. Οι καταναλωτές πρέπει να κάνουν ενημερωμένες επιλογές όταν αγοράζουν. Και εδώ ακριβώς βρίσκεται η υποστήριξη που δίδουμε στο ορατό τίμημα. Αν θα πρέπει να πάω σε ένα κατάστημα να πληρώσω 50 ευρώ πούμε, για μια μηχανή καφέ, εγώ ως καταναλωτής ενδεχομένως θα εκτιμήσω το γεγονός ότι θα ξέρω κατά πόσο πληρώνω 45 ευρώ για τη μηχανή και 5 ευρώ για την ανακύκλωση ή αν πληρώνω τέλο πάντων 35 για το μηχάνημα, για τη συσκευή για ένα όχι τόσο καλά σχεδιασμένο μηχάνημα, μια συσκευή και 15 ευρώ για την ανακύκλωση επειδή ακριβώ η συσκευή αυτή δεν είχε σχεδιαστεί καλά για ανακύκλωση και αυτήν αγοράζω. Οπότε κατά κάποιο τρόπο θεωρούμε ότι θα ήταν χρήσιμο να δίδουμε αυτό το είδος πληροφοριών στους καταναλωτές και αυτό ακριβώς επιμένουμε με αυτό το θέμα του ορατού τιμήματος και όπως είπε και ο εισηγητής σωστά οι φουσκωμένες τιμές δεν βοηθούν και κάπου θα πρέπει να υπάρχει τουλάχιστον δυνατότητα να στέλνουμε ένα μήνυμα στον καταναλωτή. Ας μην το αποκλείουμε λοιπόν. Τώρα, το θέμα των ειδικών στόχων συλλογή για τα WIP που ιδιαίτερο πρόβλημα. Κατά την άποψή μα, στην πρότασή μα ήδη ρυθμίσαμε το θέμα των συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού και εντωμεταξύ η συζήτηση είναι αρκετά εντονή σε σχέση με τον Ιδράργυρο και νομίζω ότι θα πρέπει να κάνουμε την αναθεώρηση των στόχων και να δούμε και λεπτομερώς το θέμα του Ιδραργύρου και του συγκεκριμένου στόχου συλλογής. Θα ήθελα όμως να σας ζητήσω να μας δώσετε κάποιο χρόνο εδώ, επειδή θα θέλαμε να έχουμε μια διεξοδική και προσεκτική εκτίμηση κόστους ωφέλους από τη στιγμή που θέλουμε να θέσουμε τους σωστούς ε, στόχους. Πρέπει να κάνουμε το σωστό. Το σημείο που τόνισε ο εισηγητής για τα αναρμονισμένες προδιαγραφές όσον αφορούν όσον αφορά μάλλον την ε, απεξεργασία και τη συλλογή. Αυτό αφορά και τις παλαιότερες οδηγίες, το παράρτημά τους, όπως επίσης και το τωρινό παράρτημα 1. Να πω πάντως ότι είμαστε αρκετά δεκτικοί, αρκετά ανοιχτοί για να προχωρήσουμε προς αυτή την ε, κατεύθυνση, γιατί νομίζω ότι ε, μια εξίσωση αυτών των περιεχομένων των δύο παραρτημάτων είναι κάτι το σημαντικό και ο εισηγητής παρουσιάζει μια νέα πρόταση, έναν διάμεσο στόχο δηλαδή συλλογής, κάτι το οποίο δεν έχουμε προβλέψει εμείς. Η Κομισιόν πάντως όσον αφορά τον προσωρινό στόχο συλλογής ε, θα τον ήθελε στο 45% και νομίζω ότι η Κομισιόν δεν θα ήταν διατεθειμένη για μείωση των στόχων κάτω το 65% μέχρι το, 2016. Ε, ε, Πάντως η ιδέα των ενδιάμεσων στόχων είναι κάτι το πολύ ελκυστικό και πολύ λογικό και θα ήθελα για άλλη μια φορά να τονίσω την δεκτικότητα και το ανοιχτό πνεύμα της Κομισιόν ε, για να το συζητήσει αυτό το θέμα και να το αξιολογήσουμε όπως πρέπει. Μετά, ένα άλλο θέμα, η στάθμιση της βάση υπολογισμού αντί για τη διετία ή τριετία και πάλι είμαστε ανοιχτοί, μπορούμε να το συζητήσουμε αν θέλετε κι εσείς. Απλοποίηση τώρα από τις 10 κατηγορίες στις 5. Το μήνυμα που στέλνουμε είναι και πάλι το ίδιο. Αν αυτό γίνεται χωρίς να υποβαθμιστεί η προστασία του περιβάλλοντος, χωρίς να μειωθούν οι φιλοδοξίες μας και αν χρησιμεύει στην αποφυγή περί του διοικητικού φόρτου, ευχαριστώ να το συζητήσουμε. Τέλος, ένα άλλο σημείο ίσον σημασία. η ταξινόμηση όλων των συσκευών διπλής χρήση από την αρχή συμφωνούμε ότι εδώ έχουμε να κάνουμε μια γκρίζα ζώνη που θα πρέπει να διευκρινίσουμε καλύτερα και στην πρότασή μας προτείναμε να το κάνουμε αυτό μέσω επιτροπολογίας και να επαναλάβω γιατί υποβάλαμε την πρόταση της ε, Επιτροπολογίας επειδή θεωρούμε ότι σε αυτήν την τεχνική και περίπλοκη συζήτηση ενδεχομένω να χρειαστεί να κάνουμε πολλές αναθεωρήσεις μελλοντικά αυτών των ορισμών πριν πραγματικά να φτάσει ο κόμπος στο χτένι και ενδεχομένω θα πρέπει να γίνουν διάφορες επιτροπολογίες εδώ. Αλλά η Κομισιόν βεβαίω δεν είναι αντίθετη αν ο νομοθέτης θέλει να α, θέσει διάφορα πλαίσια για την επιτροπολογία, ώστε να έχουμε μια κοινή κατεύθυνση εργασία. Ευχαριστώ πάρα πολύ, λέει ο Πρόεδρος. Ευχαριστώ. Είναι ε, περιορισμένο ο χρόνος μας. Ε, νομίζω ότι έχετε απαντήσει πολύ καλά πάντως. Ε, ακούσαμε τα βασικά σημεία. Ενδιαφέρον είναι στην μετάφραση ε, ότι ακούμε όλο και περισσότερους αγγλικούς όρους όπως το visible fee. Ε, αν κάποιος δεν ξέρει αγγλικά πάλι χαμένος είναι. Η Κομισιόν έχει τρεις ε, γλώσσες εργασίας αλλά ωραίο το ότι όλοι μιλάμε αγγλικά. Ε, ο, η συγητής έχει πάλι το λόγο, ο κύριος Πέτερλε είναι ήδη εδώ ε, και έχουμε ακόμα το θέμα της πρόληψης ε, του καρκίνου. Πρέπει να τελειώσουμε στις 6. Αγαπητέ συνάδελφε Φλόρενς, ε, έχετε να μας πείτε μερικά σοβα λόγια. Δεν ξέρω αν θα τα καταφέρω, αλλά θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συναδέλφους, να ευχαριστήσω και τον κύριο Γκρίπλερ για την καλή του συνεργασία και το προσωπικό του. Η Κάποιοι συνάδελφοι νομίζω ότι διάβασαν πράγματα στην έκθεσή μου τα οποία δεν ε, τα λέω εγώ. Εγώ δεν είπα ότι θέλουμε ότι θα έχουμε μηνιαίες εκθέσεις. Εγώ θέλω να μειώσω τι εκθέσεις, όχι να τις ε, αυξήσω σε αριθμό. Πολύ έτσι αυθόρμητα να ξεκινήσω από τα φωτοβολταϊκά. Η σχετική βιομηχανία στην Ευρώπη και στην Αμερική έχουν προτείνει μια εθελοντική συμφωνία και έχω πει ότι εγώ είμαι ικανοποιημένο με μια τέτοια εθελοντική ε, συμφωνία ε, και στο κείμενο γράφουμε ότι η Κομισιόν θα πρέπει σε τρία χρόνια να ελέγξει αν έχουν επιτευχθεί οι στόχοι. Εάν ε, όχι θα πρέπει να βρούμε κάποιο άλλο μέσο. Πάντως, ε, πιστεύω ότι είναι καλή η προσέγγιση αυτή. Μπορώ με ίσχο το κεφάλι να τη δεχτώ. Όσον αφορά το 65% δεν το πετυχαίνουμε εμείς στη χώρα μας. Ο συνάδελφος από την ε, Ιταλία είπε τι θα γίνει αν συνεχίσουμε με τον ίδιο τρόπο που, που φτάσαμε μέχρι εδώ. Θα πρέπει να κλείσουμε τα κενά και ένας ε, συντηρητικός από το Ηνωμένο Βασίλειο λέει ότι οι πολίτες δεν έχουν καταλάβει τίποτα. Ναι, στη χώρα σας έτσι είναι, διότι η πολιτική δεν έχει κάνει τίποτα. Τίποτα. Έτσι λοιπόν και ο πολίτης δεν μπορεί να παρακολουθήσει τις εξελίξεις. εάν ε, γίνει η εφαρμογή αυτών που είχαμε στην πρώτη οδηγία, όπως έγινε στην Αυστρία ή στις σκανδιναβικές χώρες, στη Δανία, ε, τότε μπορεί να μην ήμασταν, πια, ε, να μην ήμασταν στο 40%, να είχαμε φτάσει το 50-55%. Πιστεύω λοιπόν ότι θα το πετύχουμε αυτό το 65%. Έχω παρατείνει το χρονικό διάστημα αναφοράς κατά ένα χρόνο. όσον αφορά την παρατήρηση το θέμα της ε, ε, ε, διαχειρός επιλογής ή της επιλογής με μηχανήματα των ε, αποβλήτων. Ε, ναι, γνωρίζω ότι, ε, είναι, ότι υπάρχουν εδώ κάποιες θέσεις εργασίας για ε, ανθρώπους ανάπηρους που έτσι μπορούν να έχουν κάποιο εισόδημα. Κάτι τέτοιο δεν θα ήθελα σίγουρα να το, δεν θα ήθελα να το καταργήσω. Άλλο θέμα είναι... Το αν θέλουμε να ε, συμπεριλάβουμε και το εμπόριο και το εμπόριο είναι σημαντικό ε, θέμα για μένα. Εγώ προτείνω όταν κάποιος αγοράζει κάτι να επιστρέφει και ε, μια συσκευή ένα προς ένα. Πολύ μικροί έμποροι σε μικρά χωριά πολύ μικροί έμποροι σε μικρά ε, χωριά δεν έχουν χώρο για να χωρέσουν 40 τηλεοράσεις. Ε. Δεν θα ήθελα να διώξω από τα μικρά χωριά τις ε, επιχειρήσεις αυτές. Δεν θέλουμε να εκδιώξουμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. όσον αφορά τα πρότυπα. Ευχαριστώ τον κύριο Γκρίπλερ που ανέφερε ρητά ότι μας λείπουν τα πρότυπα και στην οδηγία για την διάθεση των αποβλήτων και σε άλλες οδηγίες. Υπάρχουν κενά που πρέπει να κλείσουμε, υπάρχουν παραθυράκια που πρέπει να κλείσουμε. Έχουμε τα κράτη-μέλη, έχουμε τα κέντρα συλλογής. Ε, ε, θα πρέπει να δούμε πόσα, πόσος εξοπλισμός συλλέγεται, πόσος ανακυκλώνεται και κατόπιν θα πρέπει να διαπιστώσουμε πού βρίσκονται τα κενά. Εάν δεν έχουμε τέτοιο έλεγχο, δεν θα πετύχουμε και το στόχο μας. όσον αφορά την ε, υποβολή αναφορών. Εάν δεν γίνεται αυτή σωστά, τότε δεν θα λειτουργήσει η οδηγία. Αυτό είναι το α και το ω. Ε, θα πρέπει τα κράτη-μέλη να μπορούν να πούν ότι να, εδώ, εδώ και εδώ έχουμε τα προβλήματα. Το αναφέρθηκε αυτό από τους συναδέλφους. Ε, ο συνάδελφος από τη δική μου πολιτική οικογένεια μίλησε για κίνητρα. Εδώ και 20 χρόνια συζητάμε το θέμα αυτό. η ε, πολιτική ομάδα απέναντι έχει άλλες απόψεις. Ε, ε, κάνανε προτάσεις τις οποίες εμείς απορρίψαμε, αλλά... Εγώ πιστεύω ότι μπορούμε να συζητήσουμε κίνητρα. Εάν έχετε κάποια καλή πρόταση, πολύ ευχαρίστως εδώ θα ήθελα να κλείσω. Είμαι στη διάθεσή σας, διότι φυσικά δεν μπορώ να απαντήσω σε όλα τώρα αυτή τη στιγμή. Ευχαριστώ πολύ. Ωραία. Ευχαριστώ πολύ, Καρλ Χάινς Φλόρενς. Σημαντική έκθεση αυτή στη στρατηγική για το περιβάλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουμε συγχρονίσει την έκθεση αυτή με την έκθεση ΡΟΣ. 9 Μαρτίου, 6 ε, ώρα, είναι η προθεσμία για τις Και εδώ ισχύει το ηλεκτρονικό σύστημα για την υποβολή τροπολογιών. Και φτάνουμε στο σημείο 22. Δράση κατά του καρκίνου. Ευρωπαϊκή σύμπραξη. Έχουμε εδώ εισηγητή τον Άλοης Πέτερλε. είναι και συντονιστής ε, μια ε, ομάδα που έχουμε εδώ στο Κοινοβούλιο για το θέμα αυτό. Και στο Βολιβέ βρεθήκαμε μαζί σε μια εκδήλωση με τις οργανώσεις ε, γιατρών και ασθενών. Ε, μακρηγορώ λίγο για να επικρατήσει η πρώτα ησυχία στην αίθουσα και να ξεκινήσει ο Αλόης Πέτερλε με την έκθεσή του. Φαντάζομαι ότι σε κάνα δύο λεπτά θα έχουμε ησυχάσει. Σας παρακαλώ όλους εσά που έχετε να κάνετε με τα ηλεκτρονικά απόβλητα, εγκαταλείψτε ήσυχα την αίθουσα, όσοι ενδιαφέρεστε για την πρόληψη του καρκίνου, να μείνετε εδώ. Okay, Alois Peterle hat das Wort. Άλλο Peter, λέξτε το λόγο. Ε, Αυτό το σχέδιο έκθεσης αφορά μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που εκατομμύρια πολιτών και η κοινωνία γενικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμετωπίζουν ήδη ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας πριν από χρόνια είχε προβλέψει ε, μεγάλη εξέλιξη του καρκίνου ε, και βλέπουμε σε ορισμένα κράτη πανδημία καρκίνου. Αφορά όχι μόνο τα άτομα μεγάλη ηλικία, αλλά και νέου, ακόμα και παιδιά. Παρά το γεγονό ότι γνωρίζουμε όλο και περισσότερο τον καρκίνο και παρά το γεγονό ότι η καταπολέμηση του καρκίνου έχει οργανωθεί περισσότερο, δεν μπορούμε να περιορίσουμε ε, τη σημαντική αύξηση των νέων καρκινοπαθών. Συντόμως ε, θα είναι η σοβαρότερη ασθένεια ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση που οδηγεί στους περισσότερους θανάτους. Αγαπητοί συνάδελφοι, στην αρχή της νέας θητείας μας και στην αρχή της θητείας μας, συντολής μας, όπου μας δίνονται μεγαλύτερες αρμοδιότητες, και όπου έχει χειριστεί και ο μόνιμος αντιπρόσωπος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, θα πρέπει να δούμε αυτό το πρόβλημα πολύ πιο σοβαρά. Στο παρελθόν ήδη είχαμε ε, εγκρίνει ψηφίσματα και είχαμε παροτρύνει το Συμβούλιο ε, και την Επιτροπή ε, να λάβουν μέτρη την καταπολέμηση του καρκίνου. Και είχαμε συνεργασία ψηλού επίπεδου, επίσης είχαμε ομάδα των Ευρωβουλευτών για την καταπολέμηση του καρκίνου. Τώρα λοιπόν στην αρχή της θητείας μας δεν χρειάζεται να ζητάμε στην, στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή να υιοθετούν δεσμευτικά ψηφίσματα, αλλά θα πρέπει να αναφερόμαστε στα συμπεράσματα στα οποία καταλήξαμε κατά την Σλοβενική Προεδρία. Και τώρα μπορούμε να αναφερόμαστε στην Ευρωπαϊκή Σύμπραξη για την καταπολέμηση του καρκίνου που αναφέρεται σε την έκθεση. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να σας πω στα αγγλικά, σας αναφέρω δύο συμπεράσματα. Αναγνωρίζει τη δέσμευση ε, του Κοινοβουλίου Ευρωπαϊκή Κοινότητα και των κρατών μελών ε, για την πρόληψη και την αντιμετώπιση των ε, μεγάλων μη μεταδοτικών ασθενειών με πρωτοβουλίε και ενέργηση για την πρόληψη των νόσων που επηρεάζουν θετικά τον υγιή τρόπο ζωής για παράδειγμα την αντιμετώπιση του καπνίσματος, τη σωματική άσκηση και την κατανάλωση επικίνδυνων προϊόντων. Επίσης αναγνωρίζει ε, το γεγονός ότι στον εργασιακό χώρο πολλοί είναι επιθυμένοι σε καρκινογόνες ουσίες και ε, αυτό θα, ε, πρέπει να μας οδηγήσει να περιορίσουμε στο ελάχιστο ε, τους κινδύνους καρκίνου. Επίσης στις 2 Δεκεμβρίου 2002 συνιστά τα κράτη-μέλη να εφαρμόσουν ε, ε, προγράμματα ε, εξετάσεων όλων των μορφών καρκίνου ως αποτελεσματική στρατηγική για το περιορισμό της θνησιμότητας και του κινδύνου του καρκίνου. Επανέρχομαι στη γλώσσα μου. Ε, ε, κομισία, Λοιπόν, ω προ την Επιτροπή θα ήθελα να πω ότι η ενέργεια της βασίστηκε ε, στα συμπεράσματα του Συμβουλίου και στις πολιτικές δεσμεύσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η Επιτροπή πιστεύει ότι ο τρίτον των περιπτώσεων καρκίνου μπορεί να προληφθεί αν υπάρξει υγιής τρόπο ζωής, έγκαιρη διάγνωση, σωστή πληροφόρηση κτλ. Προτείνει η Επιτροπή πολυτομεακή αντιμετώπιση ε, για αυτό το θέμα και αφορά όλους τους εμπλεκόμενους. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επίσης παρέχει τεχνική υποστήριξη σε όλους τους ενδιαφερόμενους. Αυτά ήθελα να υπογραμμίσω σχετικά με την Ευρωπαϊκή Σύμπραξη επειδή ο εκπρόσωπο τη Επιτροπή σίγουρα θα θέλει να προσθέσει ορισμένα πράγματα και να παρουσιάσει λεπτομερέστερα το σχέδιο. Το σημαντικό για μα είναι το εξή. Δεν έχουμε να κάνουμε πλέον με κλήσει, αλλά βρισκόμαστε ε, στη δράση, έχουμε δραστηριοποιηθεί. Γνωρίζουμε ότι μπορούμε να πετύχουμε πολύ περισσότερα. Είμαι πολύ ευτυχή που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει φιλόδοξου στόχου στα πλαίσια αυτή τη σύμπραξη, Δηλαδή μείωση 15% των νέων καρκινοπαθών μέχρι το 2010. Το οποίο σημαίνει ότι για 10 χρόνια 1,5% θα υπάρξει μείωση καρκινοπαθών ετησίω. Αυτή η σύμπραξη λοιπόν συμφωνεί με την υγειονομική στρατηγική που εφαρμόζουμε και καταδεικνύει τη στρατηγική προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περίοδο 2008-2014. Το ψήφισμα αυτό αναφέρεται, κάνει έκκληση ε, στην υγεία για όλους και σε όλες τις πολιτικές. Υπογραμμίζουμε τη σημασία της πρόληψης του καρκίνου. Υπό αυτό το πνεύμα λοιπόν, ο βασικός σκοπός της έκθεσης είναι να γίνονται κοινέ προσπάθειες των κρατών μελών και των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων με βάση ε, την αρχή της επικουρικότητας, ε, ώστε να έχουμε μεγαλύτερη πρόληψη για να μειωθεί ε, ο αριθμός των νέων καρκινοπαθών. Εκείνο το οποίο μας ανησυχεί είναι ότι οι χώρες επενδύουν 3% του προϋπολογισμού υγείας για την πρόληψη. Στην έκθεση αυτή αναφερόμαστε στο εξή ότι στο τρίτο του παραγράφου αναφερόμαστε στην πρόληψη. Ένα άλλο θέμα το οποίο υπογραμμίζουμε είναι οι ανισότητες. Υπάρχει αν θέλετε, ένα σιδρού παραπέτασμα μεταξύ Ανατολής και Δύσης όσον αφορά τις προοπτικές επιβίωση του καρκινοπαθούς. Επίσης υπάρχουν πολύ μεγάλες διαφορές ως προς την ένταση, την αντικατοικοποίηση των μεθόδων πρόληψης. Επίσης υπάρχουν διαφορές ε, στο θέμα αντιμετώπιση των καρκινοπαθών. Για να μην μιλήσουμε ε, ε, για τις διαφορές στην παρακολούθηση των καρκινοπαθών και στις στατιστικές για τους καρκινοπαθείς. Υπήρξε δύσκολο για ορισμένου να δεχθούν τις μεγάλες διαφορές. Δηλαδή ότι υπάρχουν διαφορές στην οργάνωση της αντιμετώπισης του καρκίνου μεταξύ κρατών ορισμένες χώρες έχουν προγράμματα αντιμετώπισης του καρκίνου και άλλες δεν έχουν στα πλαίσια της Συμφωνίας Λισαβόνας η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να υιοθετεί υποστηρικτικά μέτρα, οργανωμέ, αλλά χρειάζεται οργανωμένη προσέγγιση για να αντιμετωπίσουμε επιτυχώς τον καρκίνο. δεν μπορεί να υπάρξει ανταλλαγή των πρακτικών χωρίς να υπάρχει αλληλεπίδραση μεταξύ όλων των θεσμικών οργάνων. Ένα, μια τρίτη σημαντική αρχή είναι η σύμπραξη, η συνεργασία. Μπορούμε να πραγματοποιήσουμε τους στόχους μας ακόμα και αν δεσμεύσουμε τους πόρους μας οριζόντια και κάθετα. Προϋπόθεση όμως είναι για ε, το, τη καταπολέμηση του καρκίνου είναι κάτι το μόνιμο που πρέπει μόνιμα να υπάρχει στην ατζέντα όλων των θεσμικών οργάνων θα πρέπει να έχουμε κεφάλαια για να γίνεται έρευνα για τον καρκίνο. Και σημαντικό είναι να χρησιμοποιούνται οι γνώσεις που υπάρχουν ήδη. Κάτι το οποίο δεν γνωρίζουν όλες οι χώρες μέλη. Επίσης αναφέρει ρητά αυτή η έκθεση ότι ο υγιής τρόπος ζωής συνεισφέρει στην καταπολέμηση του καρκίνου και στην πρόληψη του καρκίνου. Μπορούμε να επηρεάσουμε την υγεία μας. Αυτό είναι γεγονός. Εκείνο το οποίο χαιρετίζουμε επίσης είναι ότι τα Υπουργεία Υγείας ε, στα κράτη-μέλη έχουν ειδικέ υπηρεσίες ε, που αφορούν τον υγιή τρόπο ζωής. Αγαπητοί συνάδελφοι, ή αντιμετωπίσουμε μια οικονομική κρίση, αντιμετωπίσουμε την κρίση των συστημάτων υγείας. Και εδώ ακόμα βλέπουμε ότι υπάρχουν οργανωμένες ομάδες ε, που χρειάζεται να αντιμετωπίσουν πολλές μορφές καρκίνου και προσπαθούν να βρουν περισσότερα κονδύλια ε, επειδή αυτός ο αγώνας για απόκτηση κεφαλαίων θα γίνεται όλο και εντονότερος, σημαντικό είναι να διαλέξουμε τη σωστή μέθοδο ε, στην προσπάθειά μας ε, καταπολέμησης του καρκίνου. Η σύμπραξη, όπως προτείνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, είναι τελικά το σωστό επίσημο πλαίσιο και αυτό πρέπει να το χαιρετήσουμε, να το υποστηρίξουμε και θα πρέπει να εφαρμόζεται ώστε να τον ευρύτερα και ώστε να τον ταχύτερα. Διότι πρόκειται για μια ενέργεια στα πλαίσια της οποίας το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να παίξει σημαντικό ρόλο. Είναι επίσης πολύ σημαντικό εμείς να παρακολουθούμε την αποτελεσματικότητα αυτών των μέτρων. Και αυτό προβλέπεται ήδη ε, στην ίδια τη σύμπραξη. Η αντιμετώπιση του καρκίνου, εστιάζοντας στην πρόληψη, απαιτεί μεγάλη πολιτική προσοχή. Αυτό δεν πρέπει να το υποστηρίζουν μόνο οι Υπουργοί Υγεία, αλλά θα πρέπει όλε οι κυβερνήσει και τα κοινοβούλια των διαφόρων κρατών μελών και οι περιφερειακέ υπηρεσίε να μα βοηθήσουν. Η σύμπραξη καλύπτει ε, τις οργανώσεις κοινωνίας των πολιτών, ομάδες πολιτών, βιομηχανίες, ε, ΜΜΕ, μέσα ε, κέντρα ερευνών κτλ θα πρέπει να προσελκύσει και τις οργανώσεις εργοδοτών και εργαζομένων. Δεν θα είναι επιτυχημένη η στρατηγική της Λισαβόνας εάν ε, δεν έχουμε υγιείς πολίτες, αν το εργατικό δυναμικό δεν είναι υγιές. Θα ήθελα καταλήγω να ευχαριστήσω τη Γραμματεία και τους συναδέλφους οι οποίοι αφιέρωσαν πολύ χρόνο και προσπάθεια και ευχαριστώ επίσης τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών για τις πρωτοβουλίες που ανέλαβαν και που περιέλαβα σε αυτό το σχέδιο έκθεσης. Ελπίζω να εγκρίνετε αυτή την έκθεση ώστε οι Ευρωπαίοι πολίτες και οι υγιείς και μη υγιείς να πούν ότι κάναμε τη δουλειά μας σε αυτό το τομέα. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Και βεβαίως προσβλέπω στη μελλοντική συνεργασία. Ευχαριστώ. Äh, Ευχαριστώ πολύ. Άλλο πέτρελε νιώθουμε το πάθος σου για το θέμα αυτό και αυτό είναι καλό. Έχουμε αρκετούς που ζήτησαν το λόγο. Η κυρία Λουκασεύσκα. Ε, Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Συμφωνώ με τον προλαλήσαντα ότι η πρόληψη του καρκίνου είναι μία από τι μεγαλύτερε προκλήσει και δυστυχώ δεν έχουμε αρκετό χρόνο για να συζητήσουμε αυτό το σοβαρό θέμα. Θα ήθελα να σα συγχαρώ, κύριε Σιγητά, για την έκθεσή σα, την οποία διάβασα με μεγάλο ενδιαφέρον. Συμφωνώ ότι υπάρχει ένα μεγάλο κενό μεταξύ Ανατολική και Δυτική Ευρώπη, μεγάλο χάσμα όσον αφορά την καταπολέμηση του καρκίνου. Εγώ έρχομαι από την Πολωνία, όπου υπάρχει ένα εθνικό πρόγραμμα καταπολέμησης του καρκίνου. Δυστυχώς όμως αυτό το πρόγραμμα ε, δεν έχει αποτελέσματα. Ε, νομίζω λοιπόν ότι ποτέ τα προγράμματα ή τα χρήματα δεν θα αλλάξουν αυτέ τι λάθο στατιστικές μεταξύ των νέων κρατών μελών, εάν εμεί δεν κάνουμε δοκιμέ, εάν ε, δεν κάνουμε εξετάσει, αν δεν πηγαίνουμε στου γιατρού, αν δεν κάνουμε τεστ. Μερικέ φορέ διστάζουμε να πάμε και σε γυναικολόγο ε, θα πρέπει να πηγαίνουν στους γιατρούς. Αλλά χρειάζεται πολλής χρόνος για να βρει κανείς ένα ραντεβού σε έναν ειδικό γιατρό. Λοιπόν, αυτό που δεν καταλαβαίνουμε είναι πόσο σημαντικό είναι να υπάρξει ένας διεθνής φορέας για την προώθηση ε, της πρόληψης ε, και για την ε, εφαρμογή των βέλτιστων πρακτικών. Σε ε, γειτονικέ χώρες υπάρχουν καταπληκτικά αποτελέσματα ναι, με μειωμένη θνησιμότητα και νοσηρότητα. Αλλά υπάρχει αυτό το κενό, αυτή η μεγάλη διαφορά μεταξύ των χωρών μας. Και βλέπουμε πόσες γυναίκες καταλήγουν καθημερινά λόγω κακής πρόληψης. Ε, και πρέπει να δούμε με βάση τι στατιστικές γιατί ορισμένε χώρες ε, επιτυγχάνουν και άλλες αποτυγχάνουν παταγωδώ. Θα ήθελα να έχω περισσότερες πληροφορίες ώστε να ετοιμαστούμε καλύτερα για να αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα καλύτερα στην Πολωνία. Στην έκθεσή σας λοιπόν Επίσης ε, υπογραμμίζετε τις εξετάσεις που γίνονται και επίσης μιλάτε για εμβολιασμό. Αλλά δεν αναφέρεται την τιμή ε, των εμβολίων, πώς θα κοστίσουν τα εμβόλια και ζείτε στις ανατολικές χώρες. Μερικές φορές πρέπει να πληρώσει κανείς 300-400 ευρώ για αυτό το εμβόλιο. Πολλές οικογένειες λοιπόν δεν μπορούν να εμβολιάσουν τις κόρες τους για καρκίνο του τραχύλου επειδή δεν έχουν τα χρήματα. Είναι πολύ ακριβό το εμβόλιο. Λοιπόν, να εστιάσουμε στη νέα γενναία, συμφωνώ. Το καλύτερο θα ήταν λοιπόν να φροντίσουμε ώστε τα νέα κορίτσια ε, πηγαίνουν στο γυναικολόγο για να κάνουν εξέταση μαστού, ότι πηγαίνουν τακτικά στον γυναικολόγο. Και πάλι ευχαριστώ πολύ και συγχαρητήρια για την έκθεσή σας κύριε Σιγητά. Ευχαριστώ η Dagmar Ροτπέρεντ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Είναι θέμα το οποίο προσπαθούμε πολλοί από εμά να το συζητήσουμε χωρίς ε, μίση και πάθη. Καταρχήν να ευχαριστήσω ε, τον εισηγητή για μια πολύ καλή έκθεση. Πιστεύω όμω επίση ότι θα έχουμε μεγαλύτερη επιτυχία εάν, να το πω έτσι, συγκεντρωθούμε. Δεν υπάρχει τίποτα λάθος στην έκθεση του Ναντίον. Ε, κάθε λέξη είναι απόλυτα σωστή, ο κύριος Πέτερλε είναι εμπειρογνώμονας. Όταν όμως ακούμε τι κάνει το Συμβούλιο και η Κομισιόν, πιστεύω ότι θα είναι καλύτερο να περιοριστούμε όχι να έχουμε 30 αιτήματα, αλλά να έχουμε πολύ συγκεκριμένα ε, αιτήματα. Ο κύριος Πέτερλε ανέφερε τι ποσοστό του προϋπολογισμού των κρατών μελών δίδεται για την πρόληψη. Ε, εγώ έχω λίγο διαφορετική προσέγγιση. Ναι, πολύ μεγάλο θέμα ε, είναι η ενημέρωση των νέων. Αλλά μεγάλο μέρος αυτού που πρέπει να κάνουμε εδώ είναι να ε, απευθύνουμε συγκεκριμένες εκκλήσεις προς τα κράτη-μέλη. Ε, συγκεκριμένες απαιτήσει να έχουμε από τα κράτη-μέλη. Ακούω για παράδειγμα ε, ότι στην ε, Πολωνία υπάρχει ένα κέντρο πρόληψης του καρκίνου. Δηλαδή υπάρχει μόνο ένα μεγάλο νοσοκομείο που να μπορεί να να υπάρχει μόνο ένα νοσοκομείο για το οποίο να μπορούν να πάνε γυναίκε με καρκίνο του μαστού και να μην ξέρουν ότι η μαστογραφία είναι ο καλύτερο τρόπο πρόληψη. Κάτι μελη που είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης πολύ περισσότερα χρόνια, όπως για παράδειγμα το Ηνωμένο Βασίλειο, κάθε δύο-τρία χρόνια καλούν τις γυναίκες να κάνουν μαστογραφία. Υπάρχουν ε, ομάδες κινδύνου στις γυναίκες για τις οποίες είναι σκανδαλώδες κάτι τέτοιο. Υπάρχουν ε, χώρες όπου δεν είναι υποχρεωτικός ο υπέρηχος για γυναίκες σε ομάδα υψηλού κινδύνου, όπως ε, για παράδειγμα οι γυναίκες που ε, είχαν ε, μαστογραφείο. Τι πρέπει να γίνει λοιπόν, να δοθούν χρήματα. Ναι, φυσικά είναι καλύτερο να δίδονται περισσότερα χρήματα. Ναι, είναι καλύτερο να εξετάζουμε τις βέλτιστες πρακτικές. Ναι. Δεν και, και τι είναι οι, οι, οι βέλτιστες πρακτικές, ε, είναι οι ίδιες οι βέλτιστες πρακτικές σε όλες τις χώρες. Στη δική μου χώρα, το νοσοκομείο στο Φλένσμπουργκ δεν ε, γνωρίζει τα ίδια πράγματα με το Σέριτε στο Βερολίνο, το μεγάλο νοσοκομείο. Ο κύριος Πέτερλε είπε ότι δεν μπορούμε να δεχτούμε τι ανισότητε που υπάρχουν μεταξύ Ανατολή και Δύση, αλλά και στο υπόλοιπο τη ε, Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχουν ανισότητε τι οποίε ε, δεν μπορούμε να δεχτούμε. Κύριε Πρόεδρε, τι μπορούμε να κάνουμε. Η προσέγγιση μου είναι πάντα ότι κάτι πρέπει να κάνουμε. Ε, τα αιτήματα στην έκθεση αυτή είναι όλα σωστά. Αλλά όταν, ε, αν τα υιοθετήσουμε αυτά στην Επιτροπή μας και στην Ολομέλεια, τι θα αλλάξει. Μάλλον να αλλάξουμε. Θα αλλάξει κάτι. Εγώ λοιπόν θα ήθελα να έχουμε μια διαφοροποίηση αναπλοκ. Δεν υπάρχει τίποτα λάθος στην έκθεση, αλλά να έχουμε ε, ένα μπλοκ το οποίο να λέει ε, τι δεν πάει καλά και ε, ένα άλλο μπλοκ που να λέει τι πρέπει να ζητήσουμε. Θα πρέπει, για παράδειγμα, να δίδονται χρήματα για την έγκαιρη, πρόληψη, για την έγκαιρη διάγνωση, για την πρόληψη, για, την, για τον εντοπισμό τάσεων τα κράτη-μέλη θα πρέπει να αναφέρουν ε, τι ποσοστό του προϋπολογισμού για την υγεία τους δίνουν πρώτον για ε, την πρόληψη του καρκίνου, ανοίγω παρένθεση, εδώ ε, συμπεριλαμβάνεται και η έγκαιρη ενημέρωση. Δεν είναι μόνο η μαστογραφία, η, η, εξέταση για, προστάτη, για καρκίνο του προστάτη ή για καρκίνο του εντέρου ναι, συμπεριλαμβάνεται και αυτό, αλλά θα πρέπει να ενημερώσουμε του ανθρώπου ότι πρέπει να το κάνουν αυτό και μάλιστα σε κάθε περιφέρεια. Στο βαθύτερο νότο τη Βαβαρία ή στην Πορτογαλία ή στην Πολωνία. Και θα πρέπει να το πούν αυτά τα, κράτα, τα κράτη-μέλη. Θέλω κάθε χρόνο να το διαβάζω αυτό. Και η εταιρική σχέση στην οποία αναφέρεται ο κύριο Πέτερλ είναι πολύ ωραία. Αυτή έχει προγραμματιστεί για το 2013. Βρισκόμαστε τώρα στο 2010. Δεν έχουν συμβεί και πολλά πράγματα. Και δεν βλέπω να δεσμεύονται ιδιαίτερα τα κράτη-μέλη να υποχρεώνονται να δεσμεύονται να συμμετάσχουν. Ε, θα πρέπει λοιπόν να έχουμε μια σειρά ετοιμάτων προ τα κράτη-μέλη και η Κομισιόν να τα μεταφέρει αυτά στο Συμβούλιο. Δηλαδή πόσα χρήματα δίνουν, πώ μπορούν να στηρίξουν τις βέλτιστες πρακτικέ. και θυμάμαι όταν μιλούσαμε για την ομοθεσία, για ε, την ε, πρόληψη για την υγεία. Α, ακούσαμε τόσα πολλά πράγματα για τις βέλτιστες ε, πρακτικές. Δεν μας ενθουσιάζουν. Δεν ήμασταν όλοι εξίσου ενθουσιασμένοι, αλλά ε, εγώ όταν ήμουν άρρωστη δεν ήξερα ότι στην Ιταλία υπάρχουν άλλες δυνατότητες ε, θεραπείας. Ε, θα ήθελα πολύ να το ήξερα αυτό. Και νομίζω ότι είμαι από τους πιο ενημερωμένου ανθρώπους. Θα πρέπει να διασφαλίσουμε να γίνονται γνωστά αυτά τα πράγματα. Είναι υποχρέωσή μας να ε, το διατυπώσουμε αυτό. Πολύ ευχαρίστως ε, θα βοηθήσω στην ε, διαμόρφωση δύο τμήματων με συγκεκριμένα αιτήματα, ώστε κάθε χρόνο να μπορούμε να ελέγχουμε τι έχει γίνει. Ευχαριστώ πολύ, Φρεντερικ Ρίς. Oui, Monsieur le Président. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πρόεδρε, θα ήθελα να σας πω ότι όταν μου ζήτησε να πάρω το λόγο, επειδή είναι και της συγγήτρια τη Ελεύθερη Ομάδα και δεν μπορούσε να βρεθεί εδώ. Συνεπώ, εγώ σα διαβιβάζω τι δικέ τη παρατηρήσει στον ε, εισηγητή. Πρώτα απ' όλα, ευχαριστώ τον εισηγητή, εξ ονόματό τη ε, και τον συγχαίρω για αυτό το σχέδιο έκθεση που καλύπτει εν πωλής όλα τα σημαντικά στοιχεία κλειδιά για την ε, αποτελεσματική αντιμετώπιση του καρκίνου πανευρωπαϊκά. Το γεγονό ότι υπογραμμίζεται η πρόληψη και ενημέρωση ε, συμφωνική κυρία Μπαρανόβα, είναι κατα... Ε, αποφασιστική σημασία. Η διάγνωση, ε, η ανείχνευση τη ασθένεια είναι πολύ σημαντικά στοιχεία, δεδομένου ότι η πρόορη διάγνωση είναι αποφασιστική σημασία για να υπάρξει αντιμετώπιση. Επίση, υπογραμμίζει και ότι απαντώντα στην ανακοίνωση Επιτροπή, η έκθεση του Κοινοβουλίου θα μπορούσε με περισσότερε λεπτομέρειε να απαντήσει στι προτάσει που έχουν γίνει σχετικά με το θέμα τη σύμπραξη που ανέφερε ο εισηγητή, η λέξη κλειδί είναι σύμπραξη, συνεργασία και πρέπει να φροντίσει ώστε η σύμπραξη να είναι αποτελεσματική και λειτουργεί πέρα από το σλόγγαν ε, στην πράξη. Μία αξιολόγηση λοιπόν τη σωστή εφαρμογή και τη ορθής λειτουργία αυτή τη σύμπραξης χρειάζεται. Επίση, η δική μνήμα ε, στα προηγούμενα προγράμματα και στρατηγικέ για την καταπολέμηση του καρκίνου σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα ήταν ίσω χρήσιμη, σύμφωνα με την κυρία Παρνανόβα, η έκθεση αξιολόγηση ε, για την σύσταση συμβουλή όσον αφορά τη διάγνωση του καρκίνου ε, μα προσφέρει πολλά διδάγματα και θα πρέπει από εκεί να αποκομίσουμε τα μέγιστα από ό,τι έχει λειτουργήσει σωστά, από ό,τι δεν έχει λειτουργήσει σωστά, ανάλογα με τα κράτη-μέλη και για το τι δεν λειτουργήσε καθόλου, ώστε να καθορίσουμε με τον καλύτερο τρόπο αυτή την ευρωπαϊκή στρατηγική για την καταπολέμηση του καρκίνου, καθώ και το, το φύλλο πορεία που θα πρέπει να ακολουθήσουμε στη σύμπραξή μα θα ήθελα να σημειώσω ορισμένα στοιχεία σε ορισμένα συγκεκριμένα θέματα, κυρίως η ανάγκη να προωθηθεί αυτή η συνεργασία στον τομέα της έρευνας, κάτι το προφανές, η αντιμετώπιση των ανισοτήτων στην υγεία και κυρίως ε, όσον αφορά τον καρκίνο για την πρόσβαση στην, ε, στις τεχνολογίες της υγείας και στην αντιμετώπιση, καθώς και να περιληφθεί η καταπολέμηση του καρκίνου σε ε, ένα γενικό λόγω συλλογισμό για τη διαχείριση και τη σωστή λειτουργία των συστημάτων υγείας λόγω του βάρους που εκπροσωπεί αυτή η νόσος ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να σε υπόψη τι μελλοντικέ προκλήσει, όπω η γύρανση του πληθυσμού. Αυτέ ήταν οι παρατηρήσει Αντώνια. Ε, στο επόμενο γύρο θα μιλήσω προσωπικά. Äh, Μπορείτε να συνεχίσετε αν θέλετε. Σύντομα. Να παραλάβω αυτά που υπόθηκαν σε σχέση με την όθηση που είπε και ο εισηγητή και η κυρία Ροντμπέρεντ και δεν είναι πρώτη φορά που το λέμε. Κάθε φορά που θίγουμε το θέμα τη Ευρώπη και τη υγεία. θέλουμε να αποδείξουμε ότι η Ευρώπη είναι παρούσα, ότι είναι ενεργή. Εγώ βεβαίω θα ήθελα να αλλάξουμε και λεξιλόγιο, να μην λέμε θα θέλαμε, συνιστώμε νύπα. Αλλά όπως είπε και η κυρία Ροτ Μπέρεντ και ο εισηγητής, υποχρέωση, υποχρεωτικός χαρακτήρας, απέτηση, απαιτητικός, δεσμευτικός και υπάρχει και συνθήκη, ωραία, πολύ ωραία. Υπάρχει η βούλησή μας και αφενός και αφετέρου η συνθήκη. Έχουμε λοιπόν αυτό το παράδοξο με στοιχεία υπάρχοντα, αμήλικτα. Ο εισηγητής ε, μίλησε για επιδημία και μάλιστα και πανδημία για φέτος, όπως είδαμε στην επιστημονική, επιστημονική φιλολογία, λέει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ότι θα αντικαταστήσει τα καρδιαγιακά νοσήματα ο καρκίνος όσον αφορά τον αριθμό των θανάτων φέτος. Υπάρχουν και διάφορα θέματα προς την Κομισιόν, όχι το Σουσιάδη αλλά τέλος πάντων, για να προχωρήσουμε πιο γρήγορα, να πω ότι το κυριότερο ζήτημα εδώ είναι ότι αυτή η σύμπραξη θα πρέπει να συνεπάρχει με το καλύτερο δυνατό τρόπο εφαρμογή όλων αυτών των πράξεων και εξάλλου αυτό θα είναι και το αντικείμενο τη γνωμοδότηση που θα έχουμε. Είναι καλό βέβαια να μιλάμε για συνεργασία και εφαρμογή των δικτύων, αλλά αυτά θα πρέπει να υλοποιηθούν στην πράξη. Εκτό από αυτά, θα ήθελα να συγχαρώ το, την συγκίτρια για το σημείο 11 Μιλήσαμε για την πρόληψη. Επειδή ένα τρίτο του καρκίνου θα μπορούσε να αποφευθεί, περιπτώσεων καρκίνου θα μπορούσε να αποφευθεί με μια υγιεινή ζωή και ένα διαφορετικό τρόπο ζωής. Να τονίσουμε λοιπόν αυτό το ζήτημα. Ένα τρίτο είναι κάτι πολύ μεγάλο ως στοιχείο Αυτά για το 11. Για το 16 επίσης να πω ότι από το 2003 ήμουνα εισηγήτρια για το σχέδιο της διάρθρωσης των ε, της και τη σχέση μεταξύ ε, περιβάλλοντος και υγείας. Στο 16 λοιπόν έχουμε όλες τις περιβαλλοντικές αιτίε των καρκίνων που υπάρχουν σήμερα. Έχουμε τη συνεχή έκθεση σε διάφορους παράγοντες βλαβερούς που επιβαρύνει την ε, επέκταση του καρκίνου. Μετά έχουμε και το, 15, το σημείο 15 και έχουμε τις επαφές με τους γιατρούς και η επιστημονική φιλολογία μας λέει ότι μέσω διαφορών τεστ, βιολογικών τεστ, θα πρέπει να τα εφαρμόσουμε ώστε να έχουμε καλύτερη διάγνωση και καλύτερη πρόγνωση και νομίζω ότι τελικά πραγματικά η καλύτερη θεραπεία ιδιαίτερα για τον καρκίνο είναι η πρόληψη βεβαίω, αλλά και η έγκυρη πρόγνωση. Ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ και ο πρόεδρος Καρίν Καρμπάχ. Μπορώ να συνεχίσω από εκεί που σταμάτησε η προλαλή σας από τη μία ε, δυσκολεύομαι λίγο διότι μου αρέσει πολύ η πρόταση της Dagmar Rockparent να κάνουμε πιο συμπαγέ στο κείμενο και να τονίσουμε κάποια θέματα. Απ' την άλλη μπαίνουμε και στον πειρασμό να προχωρήσουμε εις βάθος. Ε, ναι, ναι εγώ θα ήθελα να προχωρήσουμε εις βάθος, αλλά επί της αρχής ε, αρέσει η προσέγγιση της Dagmar. Ε, ο καρκίνος ε, δεν, ε, δεν έχει μόνο γενετικές αιτίες, οφείλεται και σε εξωτερικά παράγοντες ε, και όπως ε, στο gender mainstreaming καλό θα ήταν να έχουμε mainstreaming και στον τομέα της υγείας δηλαδή να συμπεριλάβουμε όλες αυτές ε, τις προτάσεις να σκεφτούμε την πίεση στο χώρο εργασίας την πίεση γενικά στη ζωή και το άγχος ανήκει στους παράγοντες που μπορούν να προκαλέσουν καρκίνο θα πρέπει λοιπόν στο μέλλον να φροντίσουμε να εξετάζουμε τις ε, νομοθετικές ε, προτάσεις ε, στο μέλλον μας, πρέπει να εξετάσουμε τις μελλοντικές νομοθετικές προτάσεις, να δούμε σε τι βαθμό επιδεινώνουν την υγεία του ενδιαφερομένου. Βλέπουμε ότι σε κοινωνικά στρώματα με χαμηλό εισόδημα, με, χαμηλή, με χαμηλό επίπεδο εκπαίδευσης είναι και Πολύ σημαντικότερο πρόβλημα ο καρκίνος. Θα πρέπει λοιπόν πολύ συγκεκριμένα να απευθυνόμαστε ε, σε συγκεκριμένες ομάδες ε, με όρους που να καταλαβαίνουν ώστε και τα κοινωνικά στρώματα με ε, χαμηλότερο επίπεδο μόρφωσης και χαμηλότερο εισόδημα να μπορούν να αποφελούνται από τα μέτρα αυτά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Πέτρελ έχει και πάλι το λόγο. Να δώσω πρώτα όμως το λόγο στην Κομισιόν. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ξέρω ότι έχουμε λίγα μόνο λεπτά. Θα είμαι πολύ σύντομος λοιπόν. Δεν θέλω να πω και πολλά. Επειδή ο εισηγητής παρουσίασε ένα σχέδιο γνωμοδότησης το οποίο καλωσορίζει η Κομισιόν και ε, είμαστε γνώμονες σε εσά Πρόεδρε και στον εισηγητή για αυτή την πρωτοβουλία για την σύμπραξη για τον καρκίνο. Να ενημερώσω τα μέλη ότι αυτό που έλεγε η κυρία Ροθπέρεντ όταν είχε γίνει και τίποτα από πέρσι, να σας βεβαιώσω ότι ισχύει το αντίθετο. Είχαν ένα μεγάλο φάσμα, αξιοθαύμαστο θαύμα ανταπόκριση όσον αφορά την σύμπραξη. Είχαμε οργανώσει γιατρών, νοσοκόμων, πανεπιστημιακών, εμπειρογνωμόνων, όλες τις σημαντικέ οργανώσει σε ευρωπαϊκό επίπεδο που ανταποκρίθηκαν, κάτι το οποίο δεν είχε συμβεί ποτέ παλαιότερα. Και από την Κομισιόν προσπαθούμε να πάμε λιγότερο προς τις απαιτήσει. Καταλαβαίνω αυτό που που λέγατε προηγουμένω και αναφερθήκατε στην εσωτερική, στο εσωτερικό αυτό παράδοξο και τύφαση της συνθήκης δηλαδή τις προσδοκίες και τα αιτήματα των πολιτών και την αρμοδιότητα ή την εξουσία των οργάνων της Ένωσης. Θέλουμε όμως μέσω αυτής της υπεραξής να συνεργαστούμε όλοι μας. Δεν χρειάζεται λοιπόν να περιοριστούμε στο κατά πόσο μπορούμε να εκθετήσουμε μια οδηγία ή όχι. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τη χρονική στιγμή και την συνειδητοποίηση που υπάρχει σε όλη την κοινωνία, σε όλο το φάσμα της κοινωνίας για τον καρκίνο, ώστε να κάνουμε συγκεκριμένα βήματα προόδου και αυτό ακριβώς θέλουμε να κάνουμε. Δεν ξέρω ακριβώς ποιε είναι οι τελικές λεπτομέρειες, γιατί μόνο τον επόμενο μήνα θα υποβληθεί η τελική πρόταση για τη σύμπραξη, αλλά είχαμε διάφορες συνεδριάσεις, διάφορες συναντήσεις ώστε να συμμετάσχουν οργανώσεις από κάθε τομέα και με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουμε να κάνουμε μια σημαντική συμβολή σε αυτό το τομέα. Πρόεδρε, πάντως, το τελευταίο σημείο στο οποίο θα ήθελα να αφιστήσω την προσοχή σας αφορά την ανάγκη που έχουμε για τη δική σας υποστήριξη, όχι μόνο τώρα, αλλά για τα επόμενα χρόνια και τους επόμενους μήνες ο συγητής τόνισε την ανάγκη για βιωσιμότητα, για βιώσιμη υποστήριξη και συνεχή υποστήριξη και χρηματοδότηση. Και αυτό θα το συζητήσουμε και στις νέες χρηματοοικοδομικές προοπτικές που θα έχουμε στο άμεσο μέλλον. Βεβαίως τώρα, η κύρια χρηματοδότηση για την αντιμετώπιση αυτών των θεμάτων θα πρέπει να προέρχεται από τις χώρες μέλη και τα συστήματα υγείας τους. Υπάρχουν όμως και πολλά ευρωπαϊκά εργαλεία που υπάρχουν ακριβώς για να αντιμετωπίσουν κάποιες αδικίες μιλήσαμε για τα διαφορετικά ταμεία, για τι αδικίες, μάλλον για τις ανισότητε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ανισότητε οι οποίε επηρεάζουν την οικονομική μα απόδοση. Η οικονομική κρίση θα μπορούσε να βοηθηθεί ενδεχομένω και από τι επενδύσει στον τομέα τη υγεία μέσω μια συνεχού δέσμευσης σε αυτόν τον τομέα ώστε να διασφαλίσουμε τι απαραίτητε επενδύσει και για τον καρκίνο και για άλλα θέματα υγεία και να προχωρήσουμε. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος ε, Σπέτερλε. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Κομισιόν και τους οικειώδεις εισηγητές. Διαπιστώνω μια διαφορά μεταξύ της προηγούμενης και της επόμενης θητείας του Κοινοβουλίου γιατί πράγματι τώρα έχουμε περάσει τη δράση. Και καλό να ήταν περισσότερα εδώ στο σώμα μας. Θα ήθελα λοιπόν οι προσπάθειές μας να επικεντρωθούν σε ένα καλό ορισμό της σύμπραξης αυτής και να χαράξουμε φιλόδοξους στόχους και κατευθύνσεις. Λαμβάνοντας υπόψη όλα αυτά που είπατε προηγουμένως, βλέπω έτσι κάποια αντίθεση ανάμεσα στο επίπεδο λεπτομέρειας που θέλουμε και στη συνεκτικότητα. Βλέπω ότι υπάρχουν προτάσεις και απόψεις που θέτουν φιλόδοξους στόχους όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Σύμπραξη αυτή. Και νομίζω ότι αυτή η σύμπραξη έχει λάβει πολύ θετική ανταπόκριση. Και εγώ ο ίδιος συμμετείχα στην έναρξη των δραστηριοτήτων για αυτή την υλοποίηση αυτή της ε, σύμπραξη και είδα ότι ο κόσμος πραγματικά θέλει να υπάρξει μια αλλαγή. Χρειαζόμαστε εδώ λοιπόν διαφάνεια, σαφήνεια, δέσμευση σημαντική και ουσιώδη και φιλοδοξίες. Φιλόδοξο στόχο δηλαδή για την υγεία. Μπορεί κάποια πράγματα να μην πάνε σου μακριά όσο θα θέλαμε. Όμως η αλήθεια είναι ότι όλοι θα πρέπει να μιλάμε για ένα νέο παράδειγμα. Αν θυμάστε τις ακροάσεις που είχαμε με τους υποψήφιους επιτρόπους που μιλάνε για αλλαγή στάσης και συμπεριφοράς, όχι μόνο για την ενέργεια, του περιβάλλον. Αυτή λοιπόν η, αλλαγή στάσης και συμπεριφοράς είναι κάτι το υγιές από μόνο του. Οπότε τα πράγματα θα αλλάξουν, επειδή πρέπει να αλλάξουν και εμείς θα συμμετέχουμε σε αυτήν την αλλαγή. Από τις παρεμβάσεις λοιπόν βλέπω ότι αυτά που λέω δεν αντιτάσσονται στις πεπιθήσεις σας και ότι θα με υποστηρίξετε στις προσπαθίες μου. Νομίζω ότι θα πρέπει να κάνουμε τα διαφορετικά ταμεία το καλύτερο, το βέλτιστο εργαλείο ώστε να μειωθούν οι ανισότητες. Και θα ήθελα να ζητήσω στο τέλος αυτής της πενταετούς κοινοβουλευτικής θητείας όλα τα κράτη-μέλη να έχουν εθνικά προγράμματα ανείχνευσης του καρκίνου να ευθετηθούν όλες οι συστάσεις μας και ο κώδικας για τον καρκίνο να αναθεωρηθεί ώστε και πάλι το ξαναλέω μετά από πέντε χρόνια να έχουμε στοιχεία και στατιστικές για την ανείχνευση του καρκίνου και θα χαιρόμουν ιδιαίτερα αν το 10-15% του ΑΕΠ αντί για το 3% των χωρών μελών να πήγαινε στην πρόληψη του καρκίνου. Φιλόδοξο στόχο αυτός βεβαίω, αλλά νομίζω το 3% είναι στατιστικό σφάλμα. Και επίση είμαι πεπισμένο ότι όταν η οδηγία για την διασυνοριακή περίθαλψη θα υιοθετηθεί, τότε η γνώση θα διαχυθεί και περισσότεροι θα γνωρίζουν τις δυνατότητες που υπάρχουν και την κινητικότητα τις δυνατότητες προσφέρει η κινητικότητα. Αλλά αυτό θα γίνει μόνο μέσω διάχυσης της ε, γνώσης και ανταλλαγή της. Συνάδελφοι, θα ήθελα να σας πω με χαρά και άλλα πράγματα βέβαια, αλλά νομίζω ότι συμφωνούμε στις κύριες γραμμές αυτής της έκθεσης και εύχομαι η έκθεσή μα να τύχει τη υποστήριξη όχι μόνο στην Επιτροπή μα αλλά και στην Ολομέλεια του Κοινοβουλίου. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ για αυτή τη δουλειά που έκανε. Η προθεσμία για τι τροπολογίε είναι η 12η Μαρτίου στι 12 το μεσημέρι. Θα δούμε μετά πώ θα προχωρήσουμε βεβαίω. Η ψηφοφορία θα γίνει 7 του Απρίλη στην Επιτροπή σας ευχαριστώ όλους για τη συμμετοχή σας. Λύεται η συνεδρίαση και σε δύο λεπτά θα συνεχίσουμε με τη συνάντηση των συντονιστών.